Colleagues, please Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Καλώς ορίζοντας τον Επίτροπο Αλμούνια και ευχαριστώντας τον για την εξαιρετή συνεργασία με την Επιτροπή μας τα τελευταία πενταετία. Δεν είχαμε βέβαια μαζί σας να επεξεργαστούμε πολλά νομοθετικά θέματα. Όμως η Επιτροπή μας έχει διαπιστώσει την διάθεση για συνεργασία από πλευρά σας στο ένα εκείνο θέμα που είχαμε τη συναπόφαση στον ανταγωνισμό και γι' αυτό σας ευχαριστούμε και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη συμβολή σας στην υπόθεση αυτή. Που ενισχύει έτσι τη θέση της Επιτροπής μας στην πολιτική ανταγωνισμού. Γενικά ήταν πολύ θετική η στάση απέναντι στο Κοινοβούλιο. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αλμούνια. Θέλουμε να συστήσουμε μέσα σας κάποιες από τις πρωτοβουλίες για τα της, ε, του ανταγωνισμού. Δύο πρωτοβουλίες, λευκή βίβλος για τη συγχώνευση και κανονισμός 1-2003 ο κανονισμός antitrust. Προτείνονται αλλαγές σε κάποια σημεία για τις ε, συγχωνεύσεις και θα πρέπει ο διάδοχός σας να αποφασίσει εάν θα υποβληθεί από την Επιτροπή νομοθετική πρόταση με διαβούλευση για το Κοινοβούλιο και η ανακοίνωση επιβεβαιώνει την επιτυχία της ε, διαχείρισης Μόντι και, τα και επισημαίνει κάποια σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Μια παρουσίαση περίπου 10 λεπτών και μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Είναι η τελευταία μου εμφάνιση εδώ, ενώπιον της Επιτροπής σας, από τότε που ορίστηκα Επίτροπος το 2008, 4, ε, συγγνώμη, ε, αντικατάστασα τον Πέδρο Σόλβες στην Επιτροπή Πρώτη και στη συνέχεια συνεργαστήκαμε μαζί σας στην πρώτη Επιτροπή Μπαρόσο που ήμουν αρμόδιος για τα οικονομικά και νομισματικά και στην Επιτροπή Μπαρόσο 2 για τον ανταγωνισμό. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ο διάλογός μου με το Κοινοβούλιο ήταν απολύτως καρποφόρος όσο και ενδιαφέρον. Εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να ακούω πάντα τις απόψεις σας, να ανταλλάσσω απόψεις με όλους σας και στα δύο χαρτοφυλάκια που είχα ε, θεωρούσα πάντα ότι δεν ήταν μόνο υποχρέωση ευθύνη του Επιτρόπου, αλλά και ευκαιρία για μένα να βελτιώνουμε την αμοιβαία μας ε, κατανόηση, την αντίληψη της κατάστασης, της προκλήσεις, της εναλλακτικέ και ελπίζω να ε, έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση για το διάλογο που είχαμε και το διάλογο που θα αρχίσετε με τη αντικαταστάτρια μου. Νομίζω ότι στην ίδια αυτή έφυσα πριν από πέντε χρόνια, όταν ήρθα για την ακρόασή μου, είπα ότι η πολιτική ανταγωνισμού είχε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο για να βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Αυτή η στόχη ήταν ύψιστη προτεραιότητα και προσανατόλιζαν ε, την πολιτική ανταγωνισμού και τους κανόνες καθώς επίσης και την νομοθετική μας δραστηριότητα και την πρόταση κανονισμού. Η εμπειρία μου κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας περίπου έρχεται να ενισχύσει την αντίληψη και την αίσθηση ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι βασικό μέσο για να βελτιώσουμε τις οικονομίες μας, την ανάπτυξη να είναι πιο βιώσιμη η φόρος, να δημιουργεί εμ, θέσεις εργασίας και ευημερία για τους πολίτες. Η ετήσια έκθεση ανταγωνισμού για το 2013 είναι αυτή που σας παρουσιάζω σήμερα και τονίζει το ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Όλα αυτά τα μέσα πολιτικής βοηθούν τις εταιρείες μας να είναι πιο αποτελεσματικές, πιο παραγωγικές και πιο καινοτόμες η καταπολέμηση των τραστ και ε, των καρτέλ δίνει καλύτερες υπηρεσίες και στους ε, καταναλωτές και στις επιχειρήσεις ε, για να μην εμποδίζεται είσοδος νέων εταιριών στην αγορά και να είναι θεμητός ο ανταγωνισμός. Ο έλεγχος των συγχωνεύσεων κρατεί τις αγορές ανοιχτές και αποτελεσματικές. Η πολιτική των κρατικών ενισχύσεων βοηθάει επίσης στην επίτευξη των στόχων και στην αποφυγή ε, διασπάθησης δημοσίου χρήματος και το, χρήματος των καταναλωτών. Επίσης, το βασικό μας οικονομικό εργαλείο είναι η ενιαία αγορά και θα πρέπει ε, εκεί να καταργούμε τα εσωτερικά ε, εμπόδια και φραγμούς ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης μου το 2010 τον Ιανουάριο αναφέρθηκα στους στόχους μου πιο ειδικά και επιτρέψτε μου να τους ε, υπενθυμίσω. Ενίσχυση και αναδράση των τραπεζών που είχαν πληγεί από την οικονομική κρίση στόχος μου ήταν να ξεχρονιστεί το σύστημα κρατικών ενισχύσεων και πλήρως να συμμετέχει το Κοινοβούλιο με συναπόφαση σε θέματα αποζημιώσεων ε, που έχουν προκληθεί από αθέμητο ανταγωνισμό. Επιτρέψτε μου να πω σε κάποιες λεπτομέρειες. ήταν πολύ σημαντικό καθήκον ο έλεγχος της υποστήριξης που έδωσαν τα κράτη στις τράπεζες. 110 ευρωπαϊκές τράπεζες που είναι περίπου το 25% των συνολικών ε, στοιχείων ενεργητικού έχουν λάβει κρατική ενίσχυση άμεση από την αρχή της κρίσης και μετά που ήταν τον Οκτώβριο 2008 θυμίζω για 13 από τις τράπεζες αυτές βρήκαμε ότι η υποστήριξη θα μπορούσε να δοθεί χωρίς περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις. Έχουμε ε, διαπραγματευτεί σχέδια αναδιάρθρωσης για 52 τράπεζες, ενώ 33 εκαθαρίστηκαν με τακτικό και συντεταγμένο τρόπο. Ε, ακόμα εργαζόμαστε επί 12 υποθέσεων. Αυτή η δημόσια στήριξη της τράπεζες έγινε με δύο βασικούς τρόπους. Ε, ε, ανακεφαλαιοποίηση με ενέσεις κεφαλαίου και ε, σταθεροποιητικά εργαλεία όπως ήταν εγγύησεις κτλ. Από την αρχή της κρίσης, τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι το τέλος του 2013, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έδωσαν στις τράπεζες 608 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι περίπου 5% λίγο παραπάνω του ΑΕΠ της Ένωσης. Μέχρι ε, σήμερα οι τράπεζες ε, επιστρέφουν έντοκα αυτά τα δάνεια, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος μέχρι να ανακτηθούν όλα αυτά τα κονδύλια, τα δημόσια επαναλαμβάνω που δόθηκαν για την κεφαλαίωση των τραπεζών. Για τις εγγυήσεις μέχρι το 2009 το σύνολο έφτανε στα 835 δισεκατομμύριο ευρώ, κρατικές εγγυήσεις. Έκτοτε έχει μειωθεί αυτό το ποσό και στα τέλη του περασμένου έτους είναι στα 400 περίπου δις. Υποδιπλασιάστηκε δηλαδή. Αυτές οι εγγύησεις έχουν ε, αποφέρει τέλη στα κράτη 38 δισεκατομμύρια ενώ μόνο 3 εκατομμύρια ε, από τις εγγύσεις αυτές κινητοποιήθηκαν μεταξύ 2008 και 2013. Αυτή η πολύ μεγάλη επιχείρηση τεράστια ε, είχε τρεις επιτεύγματα. Τη βιωσιμότητα των ε, διασωθησών τραπεζών χωρίς περαιτέρω άχθος για το φορολογούμενο και καθάριση των προβληματικών και ζημιογόνων τραπεζών. Επίσης, ε, η χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων περιορίστηκε στο ελάχιστο. Βέβαια, ακόμα και αν μιλάμε για ε, αστρονομικά ποσά. Και τρίτον, νομίζω ότι με επιτυχία ε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ίσους κανόνες παιχνιδιού για τις τράπεζες που δέχτηκαν ενισχύσεις και εκείνες που δεν δέχτηκαν. Ξέρετε ότι πέρυσι ενημέρωσα και αναβάθμισα τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζες ε, μειώνεται δραματικά ε, το ποσό που καταβάλουν τα κράτη. Ε, οι τράπεζες θα πρέπει να δανείζουν την πραγματική οικονομία και να μην βασίζονται στον ηθικό κίνδυνο. Ε, ε, πρέπει να θυμίσω και να τονίσω ότι και η Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκαναν ε, πολύ μεγάλη δουλειά για την Τραπεζική Ένωση και τελικά εγκρίθηκαν οι σχετικές αποφάσεις. Έρχομαι τώρα σε ένα μεγάλο στόχο δεύτερο που σας είχα αναφέρει ξεχωρισμός των κρατικών ενισχύσεων. Είχε σχεδιαστεί για να βοηθήσει κυβερνήσει να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν θέσει εργασία επικεντρωθήκαμε σε αυτά που επηρέαζαν περισσότερο την εσωτερική αγορά και οι νέοι κανόνες είναι και πιο εύκολοι και πιο απλοί στην εφαρμογή τους. Στην πράξη, εξυγχρονισμό σήμαινε ε, την έκδοση 10 νέων κατευθυντήριων γραμμών, 5 κανονισμών και 2 σημειωμάτων νότησης. Είναι βασικά αυτά για την ε, ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και βαθύτερη εσωτερική αγορά. Μεταξύ αυτών είναι ενέργεια, περιβάλλον, αεροπλοεία, έρευνα και ανάπτυξη, ε, ενίσχυση κινδύνου για τις μικρομεσαίες, ε, περιφερειακή ε, βοήθεια και ευρυζωνικότητα. Ελπίζω η επίσημη έγκριση των τελευταίων οδηγιών τις τελευταίες οδηγίες μάλλον θα έρθει σε επόμενες εβδομάδες. Είναι ορόσημο για την εξέλιξη του δικαίου ανταγωνισμού για να μπορούν οι πολίτες και οι εταιρείες να διεκδικούν την αποζημίωσή του ε, όταν πέφτουν θύματα σε παραβίαση των ε, κοινοτικών κανόνων ε, κατά των τραστ. Είναι για πρώτη φορά που γίνεται αυτή η προσπάθεια και ο ρόλος του Κοινοβουλίου ήταν πραγματικά αποφασιστικός για να συμφωνήσει με το Συμβούλιο επί του τελικού κειμένου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερω την Επιτροπή σας και τα μέλη της που συμμετείχαν άμεσα σε αυτό το εγχείρημα. Θα έρθω τώρα σε κάποιου άλλους τομείς, κάποια άλλα παραδείγματα για το πώς δημιουργήσαμε καλές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Πρώτον, το σύστημα πληρωμών τα διατραπεζικά τέλη ε, όταν ε, χρησιμοποιούμε τα ε, κάρτες, τα λεγόμενα MIFS, κοστίζουν τελικά στους καταναλωτές περίπου 10 δισεκατομμύρια ετησίως. Επίσης, οι διαφορές από χώρα σε χώρα διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και εμποδίζουν την καινοτομία. Είχαμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, πήραμε αποφάσεις για την ε, Visa Europe ε, για χρεωστικές κάρτες το 10 και πιστωτικές το 14 που μείωσαν το κόστος των τελών από 30 μέχρι 50%. Στην τελευταία απόφαση η εταιρεία ε, δήλωσε ότι επιβάλλει τα ίδια τέλη χαμηλότερα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τον καιρό διερευνούμε την υπόθεση Mastercard και Visa International. Ε, σε ό,τι αφορά τις επιγραμμικές πληρωμές και πάλι ε, προσφύγαμε κατά μιας οργάνωσης που εκπροσωπεί τον κλάδο και ονομάζεται European Payments Council, η Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμό. Έχουμε δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα διότι ε, οι αποφάσεις κατά τον καρτέλ και οι συγκεκριμένες οδήγησαν το Συμβούλιο αυτό να εγκαταλείψει ένα σύστημα το οποίο απέκλειε ανταγωνιστές από την αγορά. Χρειαζόμαστε βεβαίως ίσους κανόνες ε, παντού και νομική ε, ασφάλεια για τους οικονομικούς φορείς, ε, λογικά τέλη για τους καταναλωτές και δημιουργήσαμε και τις προϋποθέσεις για να μπουν στην αγορά και μη ε, τραπεζικά ιδρύματα. Ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι πάντα η νομοθεσία. Γι' αυτό ευχαριστώ και πάλι την Επιτροπή σας για το έργο σας στις δύο προτάσεις που σας στείλαμε, ο συνάδελφος Μισελ Μπαρνιέ και εγώ, σχετικά με αυτά τα θέματα για την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών και προσβλέπω και στην Ιταλική Προεδρία για να επιταχύνει το έργο αυτό σε επίπεδο Συμβουλίου και ή δυνατόν να έχουμε τριμερή διάλογο κατά τη διάρκεια ε, του ενεστώτος έτους. Ε, η τεχνολογία της ε, πληροφορίας και η ψηφιακή οικονομία είναι άλλα σημαντικά παραδείγματα. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω σύντομα μερικά. Δεδομένης της απουσίας γνήσιας εσωτερικής αγοράς για τη τηλεπικοινωνία πρόσφατα ε, αναθεωρήσαμε κάποιες συγχωνεύσεις, διότι Προφανώς η εσωτερική αγορά τηλεπικοινωνιών παραμένει στόχος, δεν είναι ακόμα πραγματικότητα. Γι' αυτό ε, είμαστε υποχρεωμένοι να αναλύσουμε αυτές τις συγχωνεύσεις και η ε, αγορά αναφοράς δεν ήταν η ενωμένη αναγορά αλλά η εθνική αγορά εγχώρια κάθε φορά και ε, όταν πήραμε αποφάσεις αυτές συνοδεύονταν από μέτρα πάρα πολύ αυστηρά για να μην υπάρχουν προβλήματα για τους καταναλωτές ε, ούτε για την ε, ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό. Όπως θα θυμάστε, πριν από ένα έτος και πλέον εγκρίναμε κάποιες αποφάσεις κατά τον τραστ Apple, Apple και κάποιους βασικούς εκδότες που ε, είχαν ε, στρεβλώσει στον ανταγωνισμό και στη συνέχεια ε, κάποιους κατασκευαστές smartphones, Motorola και Samsung. Άλλες μεγάλες αποφάσεις για τα πνευματικά δικαιώματα ελήφθησαν το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά το φαρμακευτικό τομέα τους παραγωγούς σήμων. Και ελπίζω αυτές οι αποφάσεις να βοήθησαν να μειωθεί η τιμή του φαρμάκου για τους ασθενείς και τους καταναλωτές και να μειωθούν γενικά τα κόστη για τα συστήματα υγείας στα κράτη-μέλη, διότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να προστατεύεται καλά η υγεία τους και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατεύουμε την υγεία των πολιτών. Να έχουμε ένα ενιαίο γενικό σύστημα καθολικό ε, υγείας και προστασίας. Στην ψηφική αγορά έχουμε προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με την ταχεία εξέλιξη των αγορών και ότι κάποιες εταιρείες ε, ε, κυριαρχούν στην αγορά και έχουν δεσπόζουσα θέση. Αυτό αφορά κυρίως ε, εταιρείε με καινοτομία και λεγόμενα smart business που πρέπει να υποστηρίξουμε για την καινοτομία, για την ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι πρόβλημα βέβαια πάντα ανταγωνισμού, αλλά πλην όμως και αυτό έχει σημασία όταν κάποιο έχει δεσπόζουσα θέση και καταχράτη. Αυτή είναι σοβαρό πρόβλημα ανταγωνισμού. Τελειώνω με μερικά λόγια για την ε, έρευνα για την υπόθεση Google που διεξάγεται αυτό το καιρό. Έχει συγκεντρώσει πολύ ενδιαφέρον από τον τύπο, ε, τον κλάδο, πολιτικούς κύκλου και το κοινοβούλιο. Βεβαίω, ο καθένα έχει δικαίωμα να έχει ε, τις απόψεις και τις θέσεις του για ζητήματα της έρευνας αυτής ή άλλα. Ε, για τη δραστηριότητα μιας τόσο σημαντικής εταιρείας παγκοσμίως όπως είναι η Google. Ωστόσο, όταν κάνουμε έρευνες για την καταπολέμηση των καρτέλ και των τραστ και να προετοιμάζουμε τις αποφάσεις, αυτά που έχουν σημασία ως επιχειρήματα είναι αυτά που έχουν θέση στην τυπική διαδικασία. Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν απέκρουσα στεναρά τις απόπειρες ε, να γίνει αυτή μια συνηθισμένη πολιτική συζήτηση. Ε, να σας ε, εξηγήσω τώρα που βρισκόμαστε. Είναι στάνταρ πρακτική μας αυτή από το άρθρο 9 και τη σχετική διαδικασία. Εάν συμφωνεί, τελικά υπάρχει μια απόφαση που δεσμεύει. Πριν το καλοκαίρι στείλαμε κάποιες επιστολές, ήταν 20 ε, εκείνοι που κατήγγυλαν ε, ε, την εταιρεία και μας έδωσαν ισχυρά επιχειρήματα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την υπόθεση. Αρχές του μήνα τα έστειλα στην εταιρεία, τα διαβίβασα για να βελτιώσει, για να απαντήσει στα παράπονα και τις καταγγελίες, να δούμε τι συνέχεια θα δώσει και αν θα διασκεδάσει τις ανησυχίες μας. Ε, εάν απαντήσει προς τη σωστή κατεύθυνση θα συνεχίσουν αυτές οι διαδικασίες βάσει του άρθρου 9 προς εξέβρεση λύσης. Άλλως, ε, το επόμενο ε, βήμα είναι να ετοιμάσουμε μία δήλωση ενστάσεων. Ανεξάρτητα από την πορεία που θα λάβει αυτή η υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα ο Επίτροπο Αρμόδιο για τον ανταγωνισμό θα πρέπει με στένο να διατηρήσει την ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα των αποφάσεών μας. Είμαστε η πιο αξιοσέβαστη παγκοσμίω αρχή ανταγωνισμού γιατί ακριβώς διαφυλάσσουμε αυτές τις αρχές σαν κόρη οφθαλμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πέτροπε. Και τώρα δίνω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς και εγώ εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αλμούνια για τη δουλειά του. Αυτονόητο νομίζω είναι και περισσότερο από αυτονόητο. Έχετε τα τελευταία πέντε χρόνια κάνει πολύ σοβαρή δουλειά θέτοντας ορόσημα πάνω από όλα και σε αυτό είμαι ευγνώμων. Έχω λοιπόν τις εξής ερωτήσεις. Ένα θέμα πολύ σημαντικό για μένα και για τους συναδέλφους βέβαια είναι αυτό της συναπόφασης του Κοινοβουλίου στα θέματα του ανταγωνισμού. Δώσατε μια όθηση κατά τη διάρκεια της ε, θητείας σας για την ε, έγκριση επί παραδείγματι της οδηγίας για την αποζημίωση με βάση τη δικασία της ε, συναπόφασης. Τώρα θα πρέπει το Κοινοβούλιο σε όλους τους τομείς, σχεδόν όλους, πέραν ορισμένων εξαιρέσεων μόνο, να συμμετέχει στις διαδικασίες με την συναπόφαση. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν γιατί δεν ε, κάνατε πιο εντατικές προσπάθειες για την επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης και κατά τη διάρκεια της αιτίας σας και τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει ώστε το Κοινοβούλιο να έχει περισσότερη συμμετοχή σε δικασίες για τη λήψη των αποφάσεων στα θέματα του ανταγωνισμού με την προσοχή Επιτροπή. Επίση, θα ήθελα εδώ να παραπέμψω όσα είπατε για την ε, ε, αντιπαράθεση με την Google και τη σχετική διαδικασία. Τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει αν δεν προλάβετε εσεί να την κλείσετε τη διαδικασία αυτή. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει διαπραγματεύσει με κάποιε παραχωρήσει από πλευρά τη Google αλλά φαίνεται και συμφωνώ σε αυτό ότι δεν εκρίθησαν επαρκείς αυτές οι παραχωρήσεις. Πιστεύετε ότι μπορείτε να είσαστε ακόμη πιο απαιτητικοί σε σχέση με την Google και νομίζετε επίσης ότι μπορεί να έχει υποβαθμιστεί, ε, εκτιμηθεί, εκτιμηθεί προς τα κάτω δηλαδή η περιπλοκότητα του θέματος αυτού. Επίσης ε, στην ιδέα για την αντιμετώπιση των ε, trust στο χώρο των καρτέλ στον χώρο των τροφίμων. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες εκτιμήσεις να μας δώσετε, γιατί είναι κάτι το οποίο βεβαίως ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην κοινή γνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλς για τα λόγια σας. Ευχαριστώ και την πολιτική σας ομάδα επίσης για την υποστήριξη και τη συνεργασία που είχα από πολλούς όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί η συναπόφαση. Το είπα στην ακρόασή μου για την οδηγία για τις ιδιωτικές αποζημιώσεις θα είναι ε, με συναπόφαση. Και έγινε. Είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Αυτό που δεν μπορώ να κάνω ούτε κανένας επίτροπος είτε για τον ανταγωνισμό ή για διάφορα θέματα γενικών καθηκόντων, δεν μπορεί με μια πρωτοβουλία του να αλλάξει τις συνθήκες. Και η συνθήκη ορίζει πάρα πολύ ξεκάθαρα ποια θέματα εμπίπτουν εκεί ε, και ποια είναι νομοθετικού χαρακτήρα και ποια έχουν διαφορετική διαδικασία από την κανονική συναπόφαση. Ε, για παράδειγμα, εάν στο μέλλον υπήρχε κάποια νομοθετική, δεν ξέρω, οποιαδήποτε πρωτοβουλία για ένα θέμα του οποίου η νομική βάση είναι αποκλειστικά το σημείο ε, ε, τη συνθήκη που μιλάει για τον ανταγωνισμό, που είναι νομίζω 101 με 108, δεν χωράει στην απόφαση, γιατί ε, είναι θέμα της συνθήκης. Ε, ελπίζω κάποια στιγμή και μακάρι να το αλλάξουμε. Εγώ είμαι υπέρ τη απόφαση παντού. Αλλά δυστυχώ η συνθήκη άλλο ορίζει. Εκείνοι που ενέκναν τη συνθήκη και την τροποποίησαν δεν μου δώσαν σημασία. Για την Google πότε θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Όταν τελειώσει η έρευνα δεν έχω ημερομηνία. Και θέλω να το πω εδώ γιατί πάντα υπάρχουν διάφορε ερμηνείε ότι κοιτάξτε ο Αλμούνια θέλει να το κλείσει πριν φύγει. Όχι. Θέλω να τελειώσει καλά και σωστά και τι σημαίνει αυτό οι χρήστες ε, της Google και εκείνοι που θέλουν να χρησιμοποιούν αυτή την πλατφόρμα για να προβάλλουν τις επαχειρηματικές τους δραστηριότητες να μπορούν να το κάνουν χωρίς εμπόδια ρεύλωση ανταγωνισμού ή ε, κατάχρηση δεσπόζουσα θέσης ή οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει, πότε θα απαντήσει η Google εγώ μπορώ να σας πω ότι αν απαντήσει κατά τη διάρκεια ε, των εβδομάδων που μου απομένουν, θα εργαστώ εγώ μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως εργάζεται από την πρώτη στιγμή και σε αυτή την περίπτωση και σε πολλές άλλες. Αν δεν απαντήσει η Google μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, προφανώς δεν θα είναι στα δικά μου χέρια. Αν κάποια στιγμή, πριν τις 31 Δεκάτου ή μετά, η αρμόδια επίτροπος ή ο αρμόδιος επίτροπος θεωρήσουν ότι δεν ανταποκρίνεται η Google στα αιτήματά μας και στις όρους και τις προϋποθέσεις, τότε θα ε, πάρει το δρόμο της η διαδικασία. Γι' αυτό που με ρωτήσετε για την Task Force για τα τρόφιμα, Food Transfer, δεν έχω πληροφόρηση. Αν τη λάβω θα σας τη διαβιβάσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές. Ο κύριος Φερνάνδης. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Δεν είχα την ευκαιρία την περασμένη θητεία να σας ε, παρακολουθήσω ως Επίτροπο, αλλά θέλω να αξιοποιήσω τη τελευταία σας εδώ εμφάνιση για να εξάρω το ρόλο σας και το έργο σας στο Σώμα των Επιτρόπων. Όπως ξέρετε, είναι περίπλοκη οικονομική κατάσταση, προέρχεται από μια χρηματοοικονομική κρίση που έφερε τις τράπεζες και το σύνολο ε, του οικονομικού τομέα ε, στο επίκεντρο των προσπαθειών ρύθμισης στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι η Ευρώπη βρήκε έναν τρόπο συνεκτικό να αντιμετωπίζει τις κρίσεις, ε, τον οποίο το στο παρελθόν. Ωστόσο, η, η φορολογούμενοι πλήρωσαν πολύ βαριά τα σπασμένα ε, της κρίσης των κακών χειρισμών και βλέπουμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή οι καταναλωτές υποφέρουν ακόμα και πλήττονται. Καθώς αποχωρούν ε, ε, τα κράτη από διάφορες συμμετοχές που έχουν. Χρειάστηκε να ε, ενισχυθεί ο χρηματοοικονομικός τομέας, δόθηκαν κρατικές ενισχύσεις, ε, αλλά είναι γεγονός ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι πιο συγκεντρωμένες από ό,τι στο παρελθόν. Εκεί διοχετεύεται κυρίως η ευρωπαϊκή αποτεμίευση και οι οικονομίες μας, αλλά είναι εμπόδιο για ε, την ανάπτυξη. Έχουν ακόμα προβλήματα ισολογισμού οι τράπεζες και ε, βλέπουμε καταστάσεις ακόμα πολύ ε, παρόμοιες με εκείνες που ζήσαμε στην αρχή της κρίσης. Λοιπόν, δεδομένης και της εμπειρίας των τελευταίων ετών, Γι' αυτό που είπατε για τις κρατικές ανισχύσεις στις τράπεζες, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια σύσταση για ε, το έργο της Επιτροπής μας ε, το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι πολύ αυστηρή η ρύθμιση ακριβώς στο τραπεζικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, για αυτό που είπατε, πριν κάνετε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Εκτός από ένα κρατος μέλος, όχι ένα ε, και περισσότερο από ένα, αλλά όχι πολλά, δεν υπάρχουν προβλήματα συγκέντρωσης των τραπεζών, των τραπεζικών ιδρυμάτων σε μια εσωτερική εγχώρια αγορά. Ηλιανική, τραπεζική κτλ. Συνεχίζει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Όταν ζεις εδώ δεν μπορείς να πας να πάρεις ε, στεγαστικό δάνειο στη Σουηδία. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει. Ε, με πολύ λίγες εξαιρέσεις λοιπόν παραμένουν σε εθνικό επίπεδο αυτά. Το, ε, το σύστημα όμως είναι ιδιαίτερα κατακαιρματισμένο. Στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι περισσότερο πιο υλοκληρωμένα, ακριβώ είναι εσωτερική αγορά και αυτό είναι το πρόβλημα. Κατά την άποψή μου είναι ένα πρόβλημα σχετικού μεγέθους σε πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες σε σχέση και σύγκριση με τράπεζες ε, εκτός Ευρώπης που είναι ανταγωνίστριες θα δούμε αυτό πώς θα λυθεί στο μέλλον το σύστημα της συγχώνευσης των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ε, κάποια στιγμή πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα επιταχυθεί. Συμφωνώ μαζί σας που ανησυχείτε για την ανυπαρξία ε, ή την χαμηλή ε, δανειοδότηση από πλευράς τραπεζών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μια πρόταση για τη μελλοντική σας δουλειά για να προχωρήσουμε νομίζω θα ήταν να μελετήσουμε ποια είναι ακριβώς τα εμπόδια έτσι ώστε τα συστήματα ε, χρηματοδότησης που ε, να είναι χωρίς τη μεσολάβηση των τραπεζών στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους που έχουν ιδέες, πρωτοβουλίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για πολλούς κλάδους της οικονομίας θα ήταν πολύ σημαντικό αν θα μπορούσαμε να ε, άρουμε τους φραγμούς και τα εμπόδια για να μπορεί να υπάρξει μια εξωτραπεζική χρηματοδότηση. Χτες είχε έρθει ο πρόεδρος Δάγκη ενώπιόν σας και δεν θέλω καθόλου να σχολιάσω τίποτα ε, ως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις δραστηριότητε της. Αλλά πιστεύω ότι η έλλειψη... Ε, Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κεφάλαια, που γιατί χαμηλή η προσπάθεια ρευσότητας, πού οφείλεται. Υπάρχει asset quality review, η αναθεώρηση για την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και, ε, και περιμένω βγουν και τα αποτελέσματα και το stress test. Και είναι πολύ σημαντικό τα επόμενα έτη όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθούν και να ελέγχουν από πάρα πολύ κοντά πώς θα επιστρέφονται τα δημόσια κονδύλια που δόθηκαν ως ενισχύσεις για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Δεν είναι επίσημες στατιστικές, είναι κάποια στοιχεία που μπορούμε να έχουμε ε, στη διάθεσή μας από δεξιά και αριστερά από την Ευρώπη, από τη δική μας δράση για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε πάση περιπτώσει πρέπει εκ του να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τις κρατικές ενισχύσεις ή με τα κρατικά χρήματα που έχουν δοθεί και εξακολουθούν να σημαίνουν ένα κίνδυνο και ένα ρίσκο για τους καταναλωτές και για τους πολίτες και τους φορολογούμενους. τέλος, αυτά τα χρόνια γίνεται μια προσπάθεια για τη ρύθμιση των χρηματαγορών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δυστυχώς δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν πριν την κρίση. Υπάρχει ακόμα ένα παρθένο έδαφος σχεδόν ανεξερεύνητο που είναι ε, οι ε, λεγόμενες ε, shadow banking, ε, παρατράπεζες. Θα πρέπει ε, να καταλάβουμε ότι εάν είναι πιο ρυθμισμένος ο επίσημος ε, τραπεζικός τομέας θα διαφύγουν κάποια κεφάλαια προς τον ανεπίσημο. Αν βάλουμε περισσότερη τάξη στα χρηματοπιστωτικά ε, κανείς όμως δεν μπορεί να προβλέψει ότι δεν θα υπάρξει κρίση στο μέλλον. Ευχαριστώ εκ μέρους του Συντηρητικού Μεταρρυθμισμού ο κύριος Μέσσερ Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και θα επανέλθω στην υπόθεση της Google. Για να ρωτήσω πώς εξηγούνται οι καθυστερήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη διερεύνηση του θέματος του Google Search και των διαφημίσεων. Εσείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχετε απορρίψει τρία εις διαφορετικές εκδόσεις ε, προσφοράς για διευθέτηση για να καταλήξετε τελικά σε μια πολύ χαμηλότερη απαιτήσεων. Πώς γυρίσατε έτσι πίσω. Υπήρξαν ε, πιέσεις από ό,τι φαίνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, από την Axel Springer να ε, να καταπολεμήσετε την Google, να την κάμψετε και τελικά αναγκαστήκατε να οπισθοδρομήσετε. Έχετε κάνει όλη τη διαδικασία που χρειάζεται με τους ε, μάρτυρες, με τη δημοσίευση των εκθέσεων κτλ. Και ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία τρία χρόνια, με τις τρεις αιτήσεις εκθέσεις δηλαδή, κάνει έκκληση για ένα καθεστώς για τον τραπεζικό τομέα, δεδομένου ότι υπάρχει ο νέος μηχανισμός εξυγίανσης για τις τράπεζες. Θα θέλω να ρωτήσω τι στάση έχετε απέναντι στις κρατικές ενισχύσεις για το θέμα της εξυγίανσης στο μέλλον και της αφαιρεγγιότητας. Ε, τι έχετε να συστήσετε για την επόμενη πενταετία εσείς. Ο κύριος Αλμούνια. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον για την περίπτωση Google και το χρονισμό. Όντως είναι μακρά η διερεύνηση. Επίσημα και τυπικά άνοιξε η υπόθεση το 2010, 30 Νοεμβρίου 2010 και σε δύο μήνες θα κλείσει τετραετία αυτή η διερεύνηση. Αλλά η έρευνα αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Εργαζόμαστε σε ένα έδαφος αχαρτογράφητο. Δεν είχε στο παρελθόν ποτέ εφαρμοστεί η νομοθεσία. η Federal Trade Commission που είναι η Αμερικανική Αρχή Ανταγωνισμού πάρα πολύ σοβαρή και αξιοσέβαστη τέλη του 2012 έκλεισε τη δική της υπόθεση κάνοντας μια τρύπα στο νερό. Εμείς θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα για να αρθούν οι φραγμοί και τα εμπόδια στον ανταγωνισμό που υπάρχουν, σε αυτό που διερευνάτε. Τι ψάχνουν δηλαδή. Έχει αλλάξει μέσα σε αυτή την τετραετία. Κάθε μήνα αλλάζει σχήμα. Δηλαδή ένα, μια κινούμενη άμμο εξετάζουμε που αλλάζει τρόπο παροχής υπηρεσιών, φέρνει νέες υπηρεσίες, νέους συνδέσμους, νέα links. Δεν είναι εύκολο. Ξεγλιστράει. Από την άλλη έχουμε επίσημες καταγγελίες και παράπονα πάρα πολλές που όσο προχωράει η έρευνα αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 επίσημες καταγγελίες δύο από τις 20 καταπίπτουν επίσημα διότι δεν απάντησαν στις επιστολές που τους στείλαμε οι ενδιαφερόμενοι πριν το καλοκαίρι, αλλά οι 18 παραμένουν πάρα πολύ ενεργές και τρέχουν. Και πρέπει να σας πω ότι από τα σχόλια που λάβαμε καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας, και ε, σχόλια όχι μόνο από τους καταγγέλλοντες αλλά και από πολλούς άλλους. Μάθαμε πολλά και βρήκαμε και κάποια στοιχεία που πρέπει να διορθωθούν ε, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες σε Google. Δεν έχει επαναπροσανατολιστεί ούτε αμφισβητηθεί η έρευνα αυτή. Ακούμε διάφορα, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, αλλά δεν ξέρουν Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να είναι εμπειρογνώμων. Εγώ όταν ανέλαβα δεν το ήξερα και χρειάστηκε να το μάθω αυτό. Δεν έχει λοιπόν αναθεωρηθεί η έρευνα αυτή. Αυτό που έγινε ήταν ότι έχει γίνει ένα βήμα παραπέρα στην έρευνα όπως έχει συμφωνηθεί. Το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση, μια ε, πρόταση δεσμεύσεων, commitments δεν ξέρω πώς λέγεται, προτάσεις δεσμεύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επόμενο βήμα γιατί έτσι ορίζει ο κανονισμό ήταν να απευθυνθούμε σε όλους αυτούς που είχαν επίσημα υποβάλει καταγγελία. Εξηγήσαμε τι φρονούμε εμείς για τις προτάσεις της Google, την τρίτη εκδοχή τους μάλιστα, γιατί οι δύο προηγούμενες είχαν απορριφθεί από τις υπηρεσίες μας. Την τρίτη εκδοχή που μας έφερε, ε, θεωρήσαμε ότι ήταν πιο θετική Τη στείλαμε στους 20 που είχαν υποβάλει τις επίσημες τους καταγγελίες και ορισμένοι από αυτούς μας απάντησαν με εμπειρικά στοιχεία και επιχειρήματα τα οποία μας οδήγησαν στη συνέχεια να ζητήσουμε από τη Google να βελτιώσει τις προτάσεις. Έτσι δουλεύουμε. Δεν έχουμε καθόλου θεωρήσει Και θέλω να ξεκαθαρίσω και το εξής. Γίνεται λόγος για πιέσεις, ξέρω εγώ, τι πιέσεις. Υπάρχουν πάντα πιέσεις. Δεν, δεν νοείται να είσαι επίτροπος ανταγωνισμού χωρίς να δέχεσαι πιέσεις. Αλλιώς ξυπνάς το πρωί ως επίτροπος ανταγωνισμού, κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και λες ένα μήνα τώρα δεν έχω λάβει καμία πίεση. Τι, τι γίνεται, τι κάνω. Αλλά για να πω στην Google ότι πρέπει να βελτιώσει τι προτάσει τη τα επιχειρήματα, δεν είναι επιχειρήματα που διάβασα στι εφημερίδε. ούτε που άκουσα σε κάποια τηλεόραση, ξέρω εγώ. Ούτε που με έχουν ε, στείλει εμένα προσωπικά σε κάποια επιστολή ή που άκουσα σε συζητήσει στο κοινοβούλιο. Όλα αυτά τα επιχειρήματα και τα στοιχεία μου τα έχουν καταθέσει ε, κάποιοι πρωταγωνιστές ε, που έχουν κάνει επίσημη καταγγελία. Και τα επιχειρήματα δεν είναι δύο παράγραφοι, είναι 50 σελίδες είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και θα δούμε πώς θα... Δώστε μου λίγο χρόνο γιατί είναι ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση για τον ανταγωνισμό. Δεν είναι μόνο αυτό το ο ανταγωνισμός, έχουμε πάρα πολλές άλλες ε, υποθέσεις. Για τη διάρκεια τώρα. Κλείνει μια τετραετία στην έρευνα και από ό,τι φαίνεται δεν έχει ολοκληρωθεί, χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο. Η Microsoft άρχισε η υπόθεση αυτή, την άρχισε ο, ο φίλος μου ο Κάλερ Βαρμίρτ, όταν ήταν επίτροπος, δεν θυμάμαι, το 97-98, κάτι τέτοιο. Η τελευταία απόφαση για τη Microsoft, για το πρόστιμο που πρότεινα στους επιτρόπους κατά της Microsoft, γιατί είχε παραβιάσει το 2009 τις αποφάσεις, 500 εκατομμύρια ήταν, δεν είναι καταφρόνητο ποσό. Αυτή η απόφαση ελήφθη λοιπόν πέρσι, το 2013, από το 97. Κοιτάξτε, μέχρι το 2013. Υπολογίστε πόσα χρόνια είναι τετραπλάσια διάρκεια από αυτή την έρευνα για την Google. Και δεν είναι και η μοναδική που θα υπάρξει για την Google, σας λέω. Θα έχουμε περισσότερες. Γιατί υπάρχουν περισσότερα προβλήματα στη λειτουργία της Google. Ακόμα και αν δεν είναι επίσημη η διαδικασία, έχει πάρει το δρόμο της. Και σε αυτή τη θητεία και οι επόμενοι που θα σας διευθύνουν στην επόμενη θητεία θα συνεχίσουν να το συζητάνε με τον αρμόδιο επίτροπο. Ευχαριστώ. Θα σας πρέπει να σας παρακαλέσω να μείνετε στα 5 λεπτά γιατί διαφορετικά δεν θα έχετε όλη τη δυνατότητα να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι λοιπόν στις ερωτήσεις σας αλλά και στις απαντήσεις σας. Επόμενος ομιλητής Παλώμα Λόπες από την ΚΟΕ. Α, όχι, με συγχωρείτε. Άλντε Μάικλ Τόιερ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς εκ μέρους της ομάδας Άλντε να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία. Έχετε ήδη τονίσει τις προσπάθειες που η Επιτροπή για ένα καλό ανταγωνισμό, για ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και από την απάντησή σας αντιλαμβανόμαστε ότι στην περίπτωση της Google μπήκατε σε χαρτογράφικτο πεδίο. Βέβαια δεν μπορεί να είναι το μόνο θέμα που θα συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή, αλλά είναι προφανές ότι η περίπτωση της Google είναι μία υπόθεση πολύ θεμελιώδους σημασίας και δεδομένου και του ε, δυναμικού συγκέντρωσης που φτάνει μέχρι το 80% έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το αντιμετωπίσουμε. Οι οικονομίες ε, του δικτύου τίνουν σε μονοπόλια και ιονή μονοπόλια έχουν όλο και μεγαλύτερη οριζόντια αλλά και, ε, εγκάρ, και κατακόρυφη συγκέντρωση και γι' αυτό πρέπει να δούμε εάν είναι επαρκές το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επαρκώς ισχυρό ώστε να προστατέψει τον καταναλωτή από αυτή την αγορά, από αυτή τη δύναμη στην αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Έχετε μπει σε χαρτογράφητο πεδίο. Βλέπετε από πλευρά σας τη δυνατότητα η νομοθεσία περί ανταγωνισμού που έχουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κριθεί επαρκής ή πιστεύετε ότι λόγω και των ε, τεχνολογικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα θα χρειαστούν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το ε, μοντέλο αγοράς που μέχρι τώρα εφαρμοζόταν μπορεί να ισχύει ακόμη ή μήπως πιστεύετε ότι θα χρειαστεί ένα διαφορετικό μοντέλο αγοράς ε, ως βάση της νέας πολιτικής για τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος. Ε, ευχαριστώ. Για την Google. Βεβαίως χρειάζεται δράση. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, όλο δράση είμαστε. Και σε αυτή την έρευνα στην οποία μπήκα σε λεπτομέρειες, αλλά προετοιμάζουμε και μια ενδεχόμενη δεύτερη έρευνα για το Android και έχουμε λάβει καταγγελίες που μας οδηγούν να διερευνήσουμε την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης για τον ανταγωνισμό η ενδεχόμενη στρέβλωση της κυκλοφορίας, δηλαδή κυριαρχία στον domain σε υπηρεσίες της Google που δεν είναι αναζήτησης, ειδικέ υπηρεσίες και αυτή είναι μια ενδεχόμενη τρίτη έρευνα βάσει του ε, άρθρου 102 της συνθήκης. Να δράσουμε μπορούμε ενδεχομένως στο μέλλον, όπως και σήμερα και με άλλες πολυεθνικές εταιρείες, αν υπάρξουν προβλήματα από πλευράς ε, καταβολής φόρων και κρατικών ενισχύσεων μας επιτρέπει το σύστημα να δράσουμε. Έχουμε αρχίσει ήδη απέναντι σε κάποιες εταιρείε και δεν αποκλείω από αυτά που διαβάζω και από αυτά που γνωρίζω στο μέλλον τέτοιου είδους δράσεις. Δεν αποκλείω, επαναλαμβάνω, ότι δεν θα αφορά την, Google. Αυτό δεν μπορώ να το ε, προεξοφλήσω. Και υπάρχουν και άλλοι τομείς που δεν είναι του ανταγωνισμού, όπως είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής που είναι και αυτό θέμα ανταγωνισμού, ε, συγγνώμη, ε, ρύθμισης. Ε, θέματα copyright, ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Ούτε αυτό μπορεί να λυθεί έτσι. Καμιά φορά, όπως είπα στην αρχή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα πνευματικά δικαιώματα ε, υπάρχουν, αλλά δεν αλλάζει έτσι η ρύθμιση μέσω μιας απόφασης ανταγωνισμού. Είναι ένα ευρύτατο πεδίο λοιπόν, το οποίο θα χρειαστεί δράση παντού σε πολλές παράλληλες λεωφόρους ή δρόμους. Εδώ βρισκόμαστε. Χρειάζεται νομοθεσία. Σας είπα δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται, όχι μόνο για την Google. Χρειάζεται νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, πιο ισχυρή από αυτή που έχουμε κατά την άποψή μου. Και επίσης χρειάζεται νομοθεσία για το copyright και τα πνευματικά δικαιώματα πιο ισχυρή από αυτή που διαθέτουμε. Και ενδεχομένως να χρειαζόταν και νομοθεσία αλλά εδώ μας περιορίζει η συνθήκη και εσάς και μας για τα θέματα τα φορολογικά. Εγώ ως πολίτης και ως πολιτικός δεν μπορώ να καταλάβω ότι έχουμε σχεδόν σηκώσει τα χέρια ψηλά όταν έχουμε φορολογικούς παραδείσους και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όχι μόνο είναι άδικο αλλά ε, στρεβλώνουν και την αγορά. Ε, δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό, δεν το καταλάβω. Όσο μου επιτρέπει το πεδίο που με αναλογεί δρώω αλλά έχω και εγώ τα όρια μου. Η Παλώμα Λόπες λοιπόν από την ΚΟΕ τώρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Όταν το κράτος δεν ρυθμίζει καλά, η αγορά ε, ε, φανερώνει ε, στρεβλώσεις. Το κράτος λοιπόν θα πρέπει να ρυθμίζει και να επιβάλλει και την τηρήση. Αυτά τα είπατε εσείς κύριε Αλμούνια το 2010 όταν κληθήκατε το κράτος ε, για τη ε, βοήθεια ε, και για τα στρεβλά της οικονομίας και τα προβλήματα που είχαμε και με τα λογιστικά και με εσφαλμένες αποφάσεις που είχαν ληφθεί και από κυβερνήσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εχθές ήμουνα στο Μπιλμπάο. Είναι θαυμάσια η χώρα των Βάσκων και είναι και η παρίδα σας. Ε, ο κόσμος ε, πλήττεται από τις εξώσεις, από καταχρηστικές ρήτρες που εφαρμόζονται στην Ισπανία και θεωρούνται απαράδεκτες ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να φορούν πάνω από ένα εκατομμύριο. Είναι κάποιες ρήτρες που έχουν επιβάλει στα δάνεια στεγαστικά κάποια, στεγαστικά, κάποιες ταμιευτήρια και τράπεζες. Ε, έχουν σωθεί από δημόσια κονδύλια αυτές οι τράπεζες στην Ισπανία. Γιατί δεν τιμωρούνται. Ε, πώς μιλάτε για ανταγωνισμό όταν μειώνονται οι μισθοί. 12,4% στην Ισπανία είναι εργαζόμενοι φτωχοί και 13% στην Ελλάδα, πάνω από 10% στην Ισπανία. Αντί να κάνετε ε, κρατικές επενδύσεις σε βιομηχανία, κρατικές ενισχύσεις ε, σώζεται ε, αυτοκινητοδρόμους με κρατικά κονδύλια. Γιατί ε, δεν προχωρήσατε στη φορολογική εναρμόνιση έτσι ώστε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και να έχουν φορολαφρήσεις και dumping εμπορικό σε κάποιες χώρες. Αυτά είναι θέματα ανταγωνισμού. Πότε αποφασίσατε να σταματήσετε να είστε κρατική λειτουργή και να ε, βάζετε τα συμφέροντα των λίγων να επικρατούν ε, και να καταπιέζουν τους πολίτες. Τα διοικητικά συμβούλια των πολυεθνικών ε, και ε, των τραπεζών ε, έχουν υποτάξει κυβερνήσεις. Δεν περιμένω να μου απαντήσετε ειλικρινά κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας διαβιβάσω τη φωνή των εργαζομένων ανδρών και γυναικών που δυστυχώς δεν γίνεται ποτέ ακουστή. Η Coca-Cola, οι γυναίκες, οι καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών από την Ελλάδα και τόσοι άλλοι. Γιατί, πού είναι όλοι αυτοί οι άνεργοι της Ευρώπης, τόσα εκατομμύρια, τι βοήθησε ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός. Αν η Ευρώπη ε, έχει καταστρεφτεί, καταστραφεί οικονομικά, κοινωνικά. Ε, τι Ευρώπη αφήνεται, φεύγεται στις 31 Οκτωβρίου. Θα τα εξηγήσετε όλα αυτά σε κάποιο βιβλίο, σε κάποιο άρθρο. Υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Στο κέντρο να είναι ο άνθρωπος. Να το κάνετε τώρα, όχι όταν φύγετε και να το πείτε και στην αντικαταστάτριά σα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που μας ενδιαφέρει να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λόπε. Πρώτον, για να μην χωράει καμιά αμφιβολία σχετικά, πέρα από τι αγωνίε σα, τι ανησυχίε σα περιγραφή των προβλημάτων για την κρίση με βρίσκουν σύμφωνο και συμπίπτουν με τη δική μου ανάλυση. Αυτό που δεν συμπίπτει με την ανάλυση μου είναι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απευθύνεστε στον κίνδυνο, η Ευρώπη. Εσείς είστε νομοθέτης. Εγώ φεύγω σε πέντε εβδομάδες, εσείς θα είστε εδώ πέντε μήνες. Βεβαίως πρέπει να γίνουν πολλά, το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει πολλά. Ορίστε, σας παρακαλώ να το κάνετε. Εξ ονόματος κυρίας Λόπες και άλλων πολλών, όλοι οι βουλευτές να κάνετε αυτά που μπορείτε να κάνετε, γιατί υπάρχει υπαρκής πλειοψηφία. Τι κάναμε εμείς. Όχι εγώ προσωπικά, αλλά η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών, όπου συζήτησε και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, την περασμένη θητεία μαζί με το, την πρωτοβουλία την νομοθετική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα είπα αυτά και τα έγραψα που είπατε, αλλά έκτοτε και μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και έχουν βελτιωθεί στη ρύθμιση των τραπεζών. Και για τις εξώσεις και τα συμπαραμαρτούντα, τι, παθαίνει κανείς όταν δεν μπορεί να πληρώσει το στεγαστικό του δάνειο. Ο Αντολίν Σάντζο Περσέδο, εξαιρετικό βουλευτή που δυστυχώ αποχώρησε, ήταν εισηγητή για μια πολύ σημαντική ε, οδηγία που ελπίζω πολύ γρήγορα να μεταφερθεί στα κράτη-μέλη. Και το ΔΕΚ απεφάνθη ε, πάρα πολύ σημαντικά κατά συγκεκριμένων εξώσεων που έχουν γίνει στην Ισπανία. Και χαίρομαι που η Ευρώπη δραστηριοποιείται σε αυτό τον κλάδο για αυτή την αδικία αλλά δεν είναι ρητορικοί οι αγώνες είναι στην πράξη με ελέγχους, με δικονομική ε, εγγύηση που είναι το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ευχαριστώ. FDD, Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Επίτροπε Αλμούνια, σίγουρα θα γνωρίζετε την κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι στην ε, χαλιβουργία του Τέρμη αυτή τη στιγμή υπήρξαν ευθύνε και δραστήριος ρόλος της ε, Τίσεν. Το επιχειρηματικό πλάνο που παρουσίασε στόχο έχει να κόψει 500 θέσεις ε, απασχόλησης στους επόμενους μήνες. Θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία εσείς αντιπροσωπεύετε είχε ε, ε, πει ότι θα εγγυηθεί αυτό το στρατηγικό τομέα όχι μόνο στην Ιταλία εγγυόμενο την ανάπτυξή του με την ασφάλεια ταυτόχρονα με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, με την προστασία του περιβάλλοντος. Υπό το φως όλων αυτών, τι θα κάνει η Κομισιόν αν τα βιομηχανικά σχέδια της Group προχωρήσει χωρίς τις αντίστοιχες επιδέσεις και με την ε, διάλυση αυτού του στρατηγικού τομέα. Τώρα, αν δούμε πως η ε, οι Γερμανοί δεν θέλουν την αύξηση της ε, νομισματικής μάζας. Πώς προτείνετε να προωθήσετε τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Χαλιβουργίας και πώς θα την προστατεύσετε από τον ε, ανταγωνισμό εκτός Ένωσης. Τώρα, στο ισοζύγιο, στο μάλλον στον ισολογισμό της εταιρείας χρειάζεται μια παρέμβαση Υποτίθεται ε, περικοπή 500 θέσεων απασχόλησης. Μήπως όμως δεν είναι ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα. Μήπως θα έπρεπε να γίνει οικονομία στα κόστη λειτουργίας και ενεργείας. Δεν είναι αυτή η λύση να κλείνουν οι επιχειρήσεις και τα εργοστάσια και να χάνονται οι θέσεις απασχόλησης. Ίσως κάτι θα πρέπει να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε από τις δικές σας αναλύσεις και αξιολογήσεις. Επίτροπε Αλμούνια, εσείς προσωπικά έχετε δεσμευτεί σε αυτή την υπόθεση που αφορά το ε, την συγκεκριμένη χαλιβουργία την Άστρια. Να μου απαντήσετε λοιπόν, όχι μόνο σε μένα, αλλά κυρίως στους 550 εργαζόμενους που σε λίγους μήνες θα χάσουν τα προστοζήν. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Επίτροπος Ανταγωνισμού προφανώς είχα την ευκαιρία επανειλημμένα να είμαι σε επαφή για την ίδια υπόθεση κατά καιρούς με την ΕΣΥΤΕ ε, που είναι το, η χαλιβουργία του Τέρνη με τις Ιταλικές αρχές, με φιλανδικές ή γερμανικές εταιρείες, με διαδικασία εξαγοράς και συγχώνευσης. Ε, δημιούργησαν πολλές εμφιβολίες ως προς το μέλλον αυτού του χαλιβουργίου. Η Οτοκούμπ, μια φιλανδική εταιρεία, αγόρασε ε, αυτή τη χαλιβουργία. Στην αρχή εμείς βάλαμε κάποιους όρους και ανταγωνισμού και προϋποθέσεις και είναι προφανές δεν μπορούν να, απελα... να είναι όλα από τα χέρια μου. Είμαι για τον ανταγωνισμό. Δεν είμαι και ο Ιταλός Υπουργό Βιομηχανίας, ούτε Κεντρική Τράπεζα, ούτε ο Επίτροπος Βιομηχανίας. Ε, εκείνο που ήταν η δική μου δουλειά ήταν ανταγωνισμός. Απευθύνθηκα λοιπόν στη φιλανδική εταιρεία και τους έβαλα μια σειρά ε, όρους και προϋποθέσεις που αντανακλώνται στην απόφαση. Τελικά γνώρισε οικονομικές δυσκολίες αυτή η φιλανδική εταιρεία και ε, επανήρθε η Thyssen Group ως κάτοχος. Και τώρα στη δεύτερη απόφαση υπάρχουν κάποιες ε, προϋποθέσεις από πλευράς ανταγωνισμού πάντα που εκ πρώτης όψεως θεωρούμε ότι τηρούνται. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν και πολλά. Αλλά σας μιλώ για τον ανταγωνισμό εγώ για να επαγρυπνούμε για το κατά πόσο και αν τηρούνται οι όροι για τη συγχώνευση. Φαίνεται ότι τηρούνται, αλλά για καλό και για κακό ε, ε, ζητήσαμε και άλλες ε, πληροφορίες και στείλαμε πολλές ερωτήσεις στους ηθήνοντες της εταιρείας οι οποίοι όταν μας απαντήσουν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή θα τα εξετάσουμε διότι θέλουμε πρώτον οι αποφάσεις μας να τηρούνται παντού και 100%. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ε, για να εγγυηθούν το μέλλον της Χαλιβουργίας Τέρνη και στις δύο μας αποφάσεις και επίσης δεν θέλουμε κανείς να χρησιμοποιεί τις δικές μας αποφάσεις ε, για ιδιωτελείς δικούς του σκοπούς που είναι εκτός πολιτικής ανταγωνισμού όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και στο συγγνώμη από τους πράσινους. Ο Μάικλ Ραϊμόν. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν Εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων δεν είμαι σε θέση ακόμα να αξιολογήσω τελικά και καταληκτικά την εργασία σας. Πολλά θέματα ακόμα θα πρέπει να κρυθούν. Θα περιοριστώ λοιπόν ε, σε ένα ζήτημα. Στο Hickle Point της Νότιας ε, Αγγλίας έχει σχεδιαστεί ένας πυρηνικός αντιδραστίας ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί αποδοτικός οικονομικά μόνο εάν διπλασιαστεί η τιμή από την κυβέρνηση του ηλεκτρικού ρεύματος σε, αυτό, σε σχέση με αυτό που είναι τώρα διαθέσιμο στην αγορά. Ε, και σας διαβάζω τώρα μία δήλωση ότι υπάρχει ο κίνδυνος ε, νέα προγράμματα καινοτόμα προγράμματα και κυρίως αυτά που μπορούν να αξιοποιήσουν ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κινδυνεύουν να τεθούν στο περιθώριο. Ε, λόγω αυτών των επιλογών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αξιολογήσει τον ε, πυρηνικό τομέα ως έναν τύπο ενέργειας ο οποίος έχει εξαντλήσει την καινοτομία του και δεν χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν είσαστε διατεθειμένος να κάνετε την έρευνα της σκοπιμότητας και της νομιμότητας πριν από την έγκριση αυτού του σχεδίου, γιατί διαφορετικά νομίζω θα αποδειχθεί το μεγαλύτερο δώρο στην βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας. Ερωτώ λοιπόν ποια είναι η δική σας θέση και τι σκοπεύετε να κάνετε. Ποια είναι η θέση σας σχέση με την πυρηνική ενέργεια πρώτα απ' όλα και τι σκοπεύετε να κάνετε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι οι αποφάσεις για το ενεργειακό μείγμα της κάθε χώρας είναι κάτι που αποφασίζουν αποκλειστικά τα κράτη-μέλη. περέστη με θερμινευόμενο. Αν αποφασίσει μια χώρα υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας, δεν είναι κάτι το οποίο περιορίζεται ή το συζητάει, το αμφισβητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το αφισβητει η ευρωπαικη όρους και το Κοινοβούλιο ε, μέχρι να αλλάξει η συνθήκη. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Αν θέλουμε να έχουμε ε, μέχρι και ενεργειακή ένωση όπως συζητείτε τώρα και είναι κάτι που ξεκίνησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη θητεία. Αυτή η αποκέντρωση τόσο σημαντικών ε, όπως είναι η πρωτογενή ε, ενέργεια και το ενεργειακό μείγμα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Εντάξει δεν είναι του παρόντος, αυτό είναι μακράς πνοής. Δεύτερο, κάθε φορά που δεχόμαστε μια κοινοποίηση για περίπτωση κρατικών ενισχύσεων, κανονικά χρησιμοποιούμε ε, τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου κλάδου. Όμως, όπως θα θυμάστε, στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον, που εγκρίθηκαν πριν από λίγους μήνες, το, την άνοιξη φέτος, αποφασίσαμε να εξαιρέσουμε, να αποκλείσουμε την πυρηνική ενέργεια από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και να αναλύσουμε τις περιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας βάσει των αρχών της συνθήκης για τον εξή απλό λόγο. Διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 18 Οκτωβρίου του 2013 δεν είχαμε λάβει κοινοποίηση που να ζητούσε να εγκρίνουμε κρατικές ενισχύσεις για πυρηνική ενέργεια. Επειδή δεν είχαμε λοιπόν προηγούμενο, ε, προτιμήσαμε να το εξαιρέσουμε από τις κατευθυντήριες γραμμές και να εξετάσουμε αυτή την αγγλική υπόθεση της 18ης δεκάτου του 13. Υπόθεση Χίνκλη. Αρχίσαμε λοιπόν μια έρευνα για να το εξετάσουμε στις 18 Δεκεμβρίου του 2013. Έκτοτε εργαζόμαστε, πρέπει να πω, με, σε αγαστή συνεργασία με τις Βρετανικές Αρχές. Εξαιρετική διαφάνεια και διάβια που θα επιθυμούσα να υπάρχει και σε άλλα θέματα. Δεν είναι η μόνη περίπλοκη περίπτωση. Εδώ υπήρχε λοιπόν δεδομένη και πολύ μεγάλη διαφάνεια και είμαστε στο παραπέντε. Θα ήθελα να υποβάλω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση απόφασης για το κατά πόσο η κρατική ενίσχυση ε, είναι συμβατή με την νομοθεσία κτλ. Πριν το τέλος της ιδίας μου ε, είναι κάποιες εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούν οι υπηρεσίες. Δεν μπορώ να σας πω ούτε την ημερομηνία ούτε να προεξοφλήσω την απόφαση γιατί είναι ακόμα στο στάδιο της εσωτερικής συζήτησης. Πρώτα θα πρέπει να σεβαστούμε τις απόψεις των υπηρεσιών Γίνεται λοιπόν αυτή η διαβούλευση μεταξύ των διαφόρων τμήματων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια με τους επιτρόπους και τα ιδιαίτερα γραφεία τους. Ευχαριστώ. τελευταία ομάδα ομιλητών θα παρακαλέσω να περιοριστεί ο καθένα σε δύο λεπτά. Θα ακούσουμε πρώτα τι ερωτήσει. Τώρα έχει μείνει λίγο χρόνο και πρέπει να αρχίσουμε το επόμενο κομμάτι τη συνεδρία σε 20 λεπτά. Ξεκινώ λοιπόν με τέσσερι ερωτήσει ομαδοποιημένε. Με τον κύριο Ροζάτη πρώτα. Δύο λεπτά. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Επίτροπε Αλμούνια, Καλώ ήρθατε και πάλι στη συνεδρίαση. Ευχαριστώ για την επικοδομητική συνεργασία που είχατε με την Επιτροπή μας και ως Επίτροπος για οικονομικά και νοσηματικά θέματα πρώτα και ως Επίτροπος Αρμόδιος για την ε, πολιτική ανταγωνισμού στη συνέχεια. Έχω τις εξής ερωτήσεις καταρχάς για την αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη που δεν είναι ακόμα ανταγωνιστική ούτε και έχει ε, δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού γιατί υπάρχουν ε, πιέσεις από εξωτερικές από εξωτερικούς ε, παρόχους φυσικού αερίου, εκ των οποίων ο πιο ε, διαβόητος για, τις, ε, για την παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού είναι η Gazprom, η οποία επιβάλλει αθέμητες τιμές σε πελάτες με συμβάσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν τη διαφοροποίηση. Επιπλέον η Gazprom αξιοποιεί ε, ε, εκμεταλλεύεται την ε, κυρίαρχη της θέση στην αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη προκειμένου να επιβάλλει τις δικές της συνθήκες για τις συμβάσεις και έτσι οι τιμές στο φυσικό αέριο παρουσιάζουν σημαντική διαφορά σε σχέση παραδείγματι με το τι πληρώνει η Λιθουανία και η Πολωνία για το φυσικό αέριο που προέρχεται από την Ρωσία που είναι κατά 50% περίπου πιο ακριβό από αυτό που πληρώνει η Γερμανία για το ίδιο φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν πρέπει να ρωτήσω εάν έχετε κάνει κάποια προσπάθεια να διερευνήσετε την συμπεριφορά της Gazprom και, μια, και επίσης να αποκαταστήσετε τον θεμητό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά φαίνεται ότι η κατάσταση είτε δεν έχει καθόλου προχωρήσει, ήταν μόνο εμβαλωματικές οι προσπάθειες. Ερωτώ λοιπόν σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε μέχρι τώρα ε, και πότε μπορούμε να δούμε την απόφαση της Επιτροπής για τα θέματα του ανταγωνισμού. Επίσης για τα... Ναι, και κοιτάξτε, ε, μια ερώτηση, έτσι φτάνει τώρα. Μιλάτε ήδη για δύο μισή λεπτά. Ναι, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι για τα τέλη ε, ενδοτραπεζικών συναλλαγών προσπαθούν να μεταφορτώσουν στον πελάτη οι τράπεζες. Έχετε δει κάποια σημάδια νομίζω τέτοιων πρακτικών. Θέλω να ρωτήσω τι πιστεύετε γι' αυτό. Υπέρβανος Περές. Αγαπητέ ε, Πίτροπε, αγαπητέ Ιωκή Μαλμούνια και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ε, θα έλεγα να σε ευχαριστήσω για τα 10 χρόνια της υποστήριξης ε, των ευρωπαϊκών ε, στόχων στο όνομα και της ομάδας μου. έχετε κάνει πολλά για την οικονομία και προσπαθήσαμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε την εμφάνιση αυτής της κρίσης που δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί. Και θα ήθελα σε αυτή την ιδιαίτερη φάση να σας θέσω δύο ερωτήσεις ε, υπό μορφή ε, απολογισμού ή διαθήκης. Καταρχήν αναφέρατε το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η πολιτική ανταγωνισμού ε, για να επαληθεύσουμε σε ποιο βαθμό Μάλλον υπό ποιου όρου επέρχεται η συναπόφαση ή ποιο είναι υπεύθυνο για το ενεργειακό μίξ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι, ποια είναι η σκέψη σας όσον αφορά το συγκεκριμένο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού. Συχνά έχω αναρωτηθεί γιατί ε, όταν πρόκειται για... Ε, ιδρύματα αξιολόγησης ε, ε, ή για ορκωτούς λογιστές κτλ. Δεν γίνονται έρευνες από πλευρά της Κομισιόν και μας, μου απάντησαν ότι δεν έχει γίνει, δεν προβλέπεται μάλλον. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Και η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την Google που είναι μια εταιρεία δυναμική σε ένα δυναμικό τομέα, καινοτόμο τομέα όπου οι Ευρωπαίοι πίστεψαν πως δεν έπρεπε πολύ να επιβάλλουμε κανόνες και ρυθμίσεις όπως ας πούμε στον τομέα της κοινωνιών ή ε, των μεταφορών. Υπάρχει όμως ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, όχι κρατικό μονοπόλιο και χωρίς καμία ρύθμιση, κανένα ρυθμιστή. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε όπως το έχουμε κάνει σε άλλες βιομηχανίες δικτύου και για το διαδίκτυο να πρέπει να σκεφτούμε κάποιον Ευρωπαίο ρυθμιστή. Σας ευχαριστώ. Γιώργος Χρήστος. Ε, με ε, κύριε Επίτροπε, έχετε πολύ καλό όνομα διεθνώς, ακόμα και στην Ελλάδα που πολλές φορές σας έχουμε κάνει κριτική, για την προσπάθειά σας να περιορίσετε τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια. Όμως, ε, θεωρώ ότι στην καθημερινή μας ζωή ε, συναντάμε συνεχώς ολιγοπόλια και μονοπόλια. Να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα και το ένα θα το ξέρετε καλά. Στην Ελλάδα είχαμε έναν κρατικό ε, αερομεταφορέα, την Ολυμπιακή Αεροπορία, Olympic Airways, την οποία επιδοτούσαμε επί σειρά ετών με δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, τέλειωσε το κρατικό μονοπόλιο. Έχουμε πάει όμως σε μια φάση ιδιωτικού ολιγοπόλιου, το οποίο δεν επιβαρύνει βέβαια τους φορολογούμενους, αλλά ανεβάζει την τιμή των εισιτηρίων πρέπει να πω ότι εσείς μας είχατε προειδοποιήσει για τους κινδύνους, δηλαδή πώς έπρεπε να οργανώσουμε την αγορά, αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι βέβαια καλύτερο από την προηγούμενη κατάσταση, δεν είναι όμως ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Ε, και ένα άλλο παράδειγμα ελληνικό. Έχουμε την ε, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, Public Power Corporation, η οποία είναι δημόσια, η οποία επιβαρύνει τους καταναλωτές, αυξάνει τα τιμολόγια αποφασίστηκε και σωστά κατά την άποψή μου να πάμε σε ένα είδος μερικής ιδιωτικοποίησης, αλλά οι πρώτες αποφάσεις πάλι έχουν σχέση με αύξηση τιμολογίων για να γίνει πιο ελκυστική ιδιωτικοποίηση και να έρθουν επενδυτές. Επομένως, σε μια χώρα που το διαθέσιμο εισόδημα έχει πέσει 25-30% υπάρχει μια γενική καχυποψία ότι μας κυβερνάνε ολιγοπόλια και μονοπόλια. Είναι τελικά ελληνική περίπτωση αυτό ή είναι μια γενικότερη τάση που ακόμα και εσείς δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Thank you. Now, Udo Ευχαριστώ, Ούντο Μπούλμαν. Κύριε Αντιπρόεδρε, και εγώ θέλω να συγχαρώ όπως και οι συνάδελφοι, το πρόσωπό σας για όλη την ε, συνεργασία και να πω ότι ε, ήταν πολύ καλά αυτά τα χρόνια και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον. Τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε το επόμενο σύντομο διάστημα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω συγκεκριμένα. Είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε στην ενιαία αγορά χωρίς μια στεναρή πολιτική για τον ανταγωνισμό. Αλλά Μήπως θα πρέπει να αναλογιστούμε και να αναδιατυπώσουμε τους όρους και τους ορισμούς της πολιτικής του ανταγωνισμού. Γιατί στην πατρίδα μου, παραδείγματι, έχουμε μικρές μεσές επιχειρήσεις οι οποίες ε, υποφέρουν από το γεγονός ότι πληρώνουν 40 με 50% φορολογία στα από της χώρας ε, με βάση την εθνική νομοθεσία ενώ άλλοι από την άλλη πλευρά των σύνορων μπορούν να πληρώνουν μέχρι και 2%. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να μιλούμε για ενιαία αγορά όταν δεν υπάρχει ε, στο θέμα της φορολογίας κάποια εξίσωση. Ίσως θα έπρεπε να αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία τύπου διαιτητικού. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ, εάν, γιατί το, και εσείς ε, κάνατε κάποια τοποθέτηση τον Ιούνιο, ε, λέγοντας ότι θέλετε να διερευνήσετε τις πρακτικές που εφαρμόζει το τομέα αυτόν. Πώς βλέπετε την, πολιτική, το μέλλον του τομέα αυτού. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Θα είμαι όσο δυνατόν σύντομος. Αλλά ήταν και πολλές ερωτήσεις. Καλώς ορίσατε και πάλι στο κοινοβούλιο. Γκάσπρομ. Τι γίνεται με την Γκάσπρομ. Ε, ανοίξαμε και επισήμω έρευνα υπό το άρθρο 102, ε, δηλαδή κατάχρηση κυρίαρχης θέσης, γιατί έχουμε καταρχήν ε, διακρίσεις στις τιμές ε, όσον αφορά τον μηχανισμό ε, τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, κατακαιρματισμός ε, της εσωτερικής αγοράς λόγω της απαγόρευσης εξαγωγής του ρωσικού φυσικού αερίου. Έπειτα, έχουμε και τις συνθήκες που συνδέονται με τα σημεία παράδοσης του ρωσικού φυσικού αερίου. Σε κάποια φάση της έρευνας, η Gazprom, οι ρωσικές αρχές δηλαδή, μας προσέγγισαν λέγοντας ας διερευνήσουμε τη δυνατότητα μιας απόφασης που θα βασίζεται σε δεσμεύσεις. Και έχουμε κάποιες αρχικές συζητήσεις επ' αυτών. Ωστόσο, όπως είπα την ε, προάλλες, στη Φλωρεντία, όπου δυστυχώς παρεξηγήθηκα, Αυτές οι συζητήσεις που στόχο έχουν την ανέβρεση πιθανής λύσης με βάση τις δεσμεύσεις σταμάτησαν όταν ξέσπασε η Ουκρανική κρίση το Μάρτιο φέτος. Όμως η έρευνα συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε και με βάση τις δεσμεύσεις με το άρθρο 9. Προχωράμε με το παραδοσιακό το διάβλο των, ε, της απαγόρευσης, άρθρο 7. Και έχουμε προχωρήσει. Και έχουμε διάφορες αντιρρήσεις λοιπόν και έχουμε προετοιμάσει μάλλον τον τοσχέ μας κατά της ΕΚΑΣΠΡΟΜ. Δεν έχει σταματήσει τελείως το πράγμα, συνεχίζεται. Ε, το είπα στην αρχική μου ομιλία. Έχουμε εδώ έναν κανονισμό τον οποίο ε, παρουσίασα μαζί με τον ε, ε, Μισελ Μπαρνιέ τον περασμένο χρόνο. Νομίζω το Συμβούλιο προχωρά τώρα πιο αργά από το Κοινοβούλιο, αλλά τώρα υπό την Ιταλική Προεδρία συνεχίζονται οι εργασίες με ταχύτερο ρυθμό. Ελπίζω πως ο τριμερής διάλογος για αυτόν τον κανονισμό θα καταστεί δυνατός πριν το τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου. Και για τις περιπτώσεις αντιτράστ έχουμε ανοιχτές για τη Mastercard ε, και την Visa International, όπου θα συνεχιστούν, αλλά και στις δύο ε, η απόφαση του δικαστηρίου, η τελική απόφαση του δικαστηρίου, που δηλώνει πως η μύψη είναι ε, αντιανταγωνιστική και ο νέος κανονισμός θα μας βοηθήσει επιτέλους να λύσουμε τα προβλήματα, διότι το να χρησιμοποιούμε το antitrust όταν έχουμε να κάνουμε τη μια φορά με τη Visa Europe, την άλλη με τη Visa International, την παράλληλη με τη Mastercard, είναι δύσκολο να τετραγωνίσει κανείς τον κύκλο. Κανονισμός συν απόφαση του ε, δικαστηρίου είναι καλή λύση. Περβάνω, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γιατί δεν ξεκινήσαμε συζήτηση υποθέσεις, οι επίσημες έρευνες με τις ε, ε, εταιρείε ε, ορκωτών λογιστών ή με τις, τα ιδρύματα αξιολόγησης, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Γιατί δεν υπάρχουν, υπάρχουν μάλλον κανονισμοί και στις δύο περιπτώσεις και ελπίζω πως θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού κατά την γνώμη μας, διότι αυτού του είδους υπηρεσία ε, τόσο τα ιδρύματα αξιολόγηση όσο και οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείε δεν ενδιαφέρονται για την σύμπτωση συμφερόντων. Θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Υπάρχει λοιπόν σοβαρό πρόβλημα ανταγωνισμού και στις δύο περιπτώσεις, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού ξεκάθαρα. Ε, μέχρι στιγμής. Ε, αν χρειαστεί βέβαια θα ενεργήσουμε. Τώρα, ρυθμίσεις για το Google και το ίντερνετ γενικότερα. Ναι, μα τι. Τι πρέπει να ρυθμίσει κανείς. Έχει κάνει την απάντηση. Γιατί εγώ έχω θέσει την ερώτηση αυτή πολλές φορές ε, όλα αυτά τα χρόνια και στον κύριο Πελερά στην Φλερ Πελερά που ήταν υπεύθυνη της διεύθυνσης, της οικονομικής διεύθυνσης ναι, ε, να μιλήσαμε για τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν για το Ιντερνετ και ρώτησα τι πιστεύετε ότι πρέπει να ρυθμίσουμε κυρία Υπουργέ. Δεν έλαβα καθαρή απάντηση. Μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει ρυθμίση στο μέλλον, αλλά σήμερα δεν ξέρω ποια, ε, ποια, είναι, ποια είναι τα στοιχεία μιας τέτοιας ε, νομοθεσίας. Και πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο του να σκοτώσουμε, να στραγγαλίσουμε την κοινοτομία σε αυτό το τομέα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ακούσαμε διάφορες προτάσεις στην Google, όχι στην έρευνα, αλλά στη δημόσια συζήτηση. Για την υπόθεση της Google άκουσα κάποιες προτάσεις Κάποιος που παρακολουθεί αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες γίνεται κατεβαίνουν ε, διαδηλωτές στο δρόμο και μας ρωτούν γιατί να στραγγαλίσετε μια υπηρεσία που είναι εξαιρετικά χρήσιμη για μας. Πρέπει όλα αυτά να τα προσέξουμε πολύ. Κύριε, Κίρτσε, κύριε Κίρτσο, Ολυμπιακή, ναι, θα πρέπει να σας θυμίσω δύο βασικές αποφάσεις. Πρώτη, Olympic Agent, ήταν αρνητική απάντηση. Δεν έπρεπε την πρώτη συγχώνευση με την Aegean. Και αργότερα οι, ίδια ίδιε εταιρείε ήρθαν, ιδιαίτερα η Aegean, και ήρθε και μου είπε: Θέλω να ξαναζητήσω μια θετική απόφαση, γιατί η Olympic πτώχευσε. Η Ολυμπιακή με πτώχευσε. Και δεν ήταν τα δικά μου λόγια αυτά, ήταν τα δικά τους. Και χρησιμοποιήσαμε εδώ στη δεύτερη θετική απόφαση την ε, πτώχευση που λέει ότι αν δηλαδή σε μια συγχώνευση η συγχώνευση δεν προχωρά θετικά και η μια εταιρεία θα εξαφανιστεί ούτως ή άλλως μπορεί να εγκριθεί η συγχώνευση γιατί το πρόβλημα του ανταγωνισμού δεν υφίσταται πλέον. Ε, υπάρχουν προβλήματα ολιγοπολίου στην Ελλάδα μάλιστα και για ορισμένες διαδρομές ναι. Ακόμα και μονοπόλιο μπορεί να πει κανείς επικρατεί. Ένα πρώην μέλος αυτού του κοινοβουλίου. Ο κύριος Κλίντς πάντα μου θυμίζει πως υπάρχει μονοπόλιο στο διαδρομή Βρυξέλλες-Φραγκφούρτο. Και εγώ, και εγώ την πατάω εκεί πολλές φορές, αλλά είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι για ποιος θα έρθει να σπάσει το μονοπόλιο. Γιατί η αρχή ανταγωνισμού θα πρέπει να ζητήσει από τους συνομιλητές της υπάρχουν φραγμοί για να έρθουν καινούργοι. Όχι, δεν υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ελπίζω πως όταν η ελληνική οικονομία θα βελτιωθεί, θα υπάρξουν νέοι, νέες εταιρείες, γιατί θα πιστέψουν ότι θα έχουν δουλειά και θα αναγκάσουν και τους άλλους να χαμηλώσουν τις τιμές τους. Ηλεκτρισμός. Τομέας ε, υπάρχει ρυθμιστής για την ενέργεια. Ναι πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι ρυθμιστές της αγοράς ηλεκτρισμού. Ε, από καιρού εις καιρό να έχουμε και περιπτώσεις αντιτράστα. Τώρα έχουμε να κάνουμε με κάποιες υποθέσεις στον τομέα του ηλεκτρισμού, πολύ σημαντικές. Αλλά λάβαμε μια πρόσφατη απόφαση από το δικαστήριο σε σχέση με μια άλλη ε, ε, ε, ελληνική επιχείρηση, τους Λιγνίτες της ΔΕΗ που έλεγε ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα που δίνονται σε μια εταιρεία δεν είναι συμβατή, συμβατά με τους κανόνες ανταγωνισμού. Πολύ σημαντική απόβαση και αυτή ισχύει και για την Ελλάδα. Και τέλος, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Φόρη, Ανέφερα προηγουμένως ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τη φορολόγηση και ε, το πρόβλημα έχει ε, και όνομα. Ομοφωνία. Θυμάμαι, όταν πήγαινα κάθε μήνα στο ΕΚΟΦΗΝ, ο συνάδελφός μου εκείνη την περίοδο, ο Λάσλο πήγαινε να συζητήσει το θέμα τη φορολογία. Σε πέντε λεπτά είχε τελειώσει, ξεπερδέψει, γιατί ένα κράτο μέλο έλεγε «Όχι, είμαι κατά». Τέλος. Δεν μπορούσαν να λάβουν απόφαση, γιατί χρειαζόταν η ομοφωνία. Και αυτή η προϋπόθεση, αυτός ο όρος της ε, ομοφωνίας δίνει λαβή για κάθε είδους κατάχρηση, εκβιασμούς και ούτω καθεξής. Και πρέπει να αντιδράσουμε, έχουμε κάποια μέσα, αλλά οι κυβερνήσεις και το κοινοβούλιο το ξέρει αυτό, μπορεί να πει, έχει λόγο, όχι μόνο η Κομισιόν να μιλήσει στις κυβερνήσεις, αλλά και το Κοινοβούλιο. Οι κυβερνήσει θα πρέπει να ξεπεράσουν τις ρητορικέ τους δηλώσεις που τις ακούσαμε τα την τελευταία φορά στα G20 στην Αυστραλία. Ε, και πρέπει να αναλύσουν την κατάσταση για να ακολουθήσουν τις συστάσεις του ΩΣΑ με ισχυρή δηλαδή ευρωπαϊκή συμμετοχή και να μπορέσουν να ληφθούν αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές δεν θα ληφθούν ούτε πρόκειται να καταλήξουν αυτές χωρίς ε, νομοθεσία και γνωρίζετε στο Κοινοβούλιο πόσο δύσκολο είναι σε αυτή τη φάση να νομοθετήσει η Ένωση επί φορολογικών θεμάτων. Σας ευχαριστώ. Τελευταία ομάδα ομιλητών τώρα. Έχετε δύο λεπτά έκαστος. Νίτερ ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας επανέλθω σε αυτό το θέμα για τις ε, πιστοτικές κάρτες γιατί δεν με έπεισε η απάντησή σας. Φαντάζομαι πως δεν χρειάζεται να ρυθμίζουμε όλα όσα θα μπορούσαν να ρυθμιστούν. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχέση κόστους ωφέλειας. Οπότε καταρχήν θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για το κατά πόσο είστε βέβαιος πως το κόστος που προκύπτει από την εισαγωγή νέων κανονισμών και επιβολή αυτών μήπως ξεπερνά τα ωφέλη, ιδιαίτερα όταν είναι σαφές ότι για τον τελευταίο ε, πελάτη, τον τελικό πελάτη, δηλαδή τον λιανοπολιτή, δεν πρόκειται αυτό να επιφέρει όφελος. Η υπηρεσία θα είναι ακριβότερη τελικά. Επίσης να ρωτήσω αν πιστεύετε πως υπάρχει πιθανότητα αυτορύθμισης σε αυτό το τομέα ή ρύθμιση μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας, ιδιαίτερα μετά από την νίκη στο δικαστήριο όπου έχουμε τα τέλη τα διατραπεζικά ε, τέλη να καλύπτονται σε κάποιους τομείς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ε, Επίτροπε, για το σπουδαίο έργο σας, λέει ο κύριος Κόφοντ. αν ε, η Κομισιόν δαπανούσε την, τα ίδια χρήματα και την, τους ίδιους πόρους ανθρώπινους και δυναμικό για την επίλυση του προβλήματος ανεργίας όπως για να συζητήσω τις τράπεζες ε, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει τώρα ε, το Περιφερικό Ταμείο πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθούν προγράμματα από το μία χώρα και από την άλλη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ε, ε, θέμη του ανταγωνισμού και τονίζουν ένα στοιχείο, ένα πρόβλημα. Πώς θα είμαστε βέβαιοι πώς το δημόσιο χρήμα θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και όχι για να μετακινούνται οι θέσεις απασχόλησης από το ένα κράτος στο άλλο. Πιστεύω πως εσείς και ο διαδοχός σας ως Επίτροπος Ανταγωνισμού θα, να, θα ε, μπορείτε να παίξετε σημαντικό ρόλο σε αυτό το τομέα και η ευθύνη για τα ταμεία ε, δεν βαραίνει μόνο εσάς, αλλά σίγουρα ως Επίτροπος Ανταγωνισμού είναι σημαντικό να εξετάσετε αυτά τα κονδύλια για να δείτε πόσο άδικα κατανέμονται, ε, ανακατανέμονται οι θέσεις απασχόληση στην Ευρώπη. Ως Επίτροπος λοιπόν Ανταγωνισμού, τι βήματα θα αναλάβετε για να καταπολεμήσετε αυτή την πρακτική και τι ακόμα βήματα μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ανδρέας Σβάμπ. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε Αλμούνια, χαίρομαι ιδιαίτερα για την καλή συνεργασία που είχαμε στην εκθέση Λουσάνου και είχαμε πολύ καλή συνεργασία σε αυτό όντως. Είναι ένα θέμα περίπλοκο και νομίζω ότι είναι ανάγκη να βρεθεί μια πρακτική και αποτελεσματική λύση. Βέβαια πρέπει να δούμε και τα κράτη-μέλη τι στάση θα τηρήσουν οι κυβερνήσεις τους και πώς ε, μπορεί να παρακολουθεί το θέμα είναι επιτροπός. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Για τον Google είπατε κάποια ενδιαφέροντα. Και γι' αυτό θέλω να σταθώ σε κάποιες πιο συγκεκριμένα σημεία. Είπατε ότι δεν μπορεί να υποτάσσεται στι εξωτερικέ πιέσει ο Επίτροπο και ότι λαμβάνει τι αποφάσει των εξαρτήτω. Ναι, αλλά παρόλα αυτά η γνώμη και η αξιοπιστία των προτάσεων στι οποίε καταλήγεται πάλι με αυτά θα κρυθεί. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω εάν ε, είχατε την ε, σκέψη να θέσετε σε λειτουργία το μηχανισμό του άρθρου 7 γιατί ανέφερε και η συνάδελφος Πέρβανς Μπερές το θέμα του, της πρακτικής εφαρμογής των διατάξεων. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αυτή τη συγκεκριμένη διάσταση και πάλι να ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία. Η κυρία Καϊλή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Επίτροπε, είναι αλήθεια πως αναλάβατε μια δύσκολη αποστολή εν μέσω μιας πρωτόγνωρης κρίσης που βρήκε απροετοίμαστη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ήταν η κρίση αυτή και μια ευκαιρία για νέες πολιτικές και μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Στρέφοντα λοιπόν την πολιτική ανταγωνιστικότητα από εκεί που ήταν κομμένη και ραμμένη για τι μεγάλε εταιρείε, θα μπορούσε να στηριχθεί με μια διαφορετική πολιτική η πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι όμως οι τράπεζες δεν δανείζουν ακόμα τις μικρές επιχειρήσεις. Σε συνθήκες δραματική ανεργία και με πολύ χαμηλού μισθού δεν έχουν πέσει οι τιμέ, ούτε έχει βοηθηθεί η οικονομική αποδοτικότητα και ενώ οι απαγορεύσεις ε, κρατικών ενισχύσεων σε κλάδους ε, που γνωρίζετε ότι απέδιδαν και δημιουργούσαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπως τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, τα δίκτυα μεταφορών, όχι μόνο δεν απελευθέρωσαν τελικά, όπως είχε προβλεφθεί, νέες δυναμικές, ε, τις δυναμικές δηλαδή των αγορών, γύρισαν τις χώρες, κυρίως του Νότου, πολλά χρόνια πίσω. Ήθελα λοιπόν να μας απαντήσετε αν πιστεύετε πως φταίνε οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ή η ίδια η φύση, ο χαρακτήρας των μεταρρυθμίσεων. Επίσης, α, όπως είπε ο κύριος Μπούλμαν, η εξίσωση στη φορολογία για μια ενιαία αγορά θα μπορούσε να γίνει πάνω σε μια στρατηγική από όλε τι χώρε κράτη-μέλη. Σε τι θα μπορούσαμε και εμεί να βοηθήσουμε πάνω σε αυτό, καθώ καταλάβαμε ότι αντιμετωπίζεται πολλά προβλήματα από τι ίδιε χώρε και ήθελα να ρωτήσω αν η στήριξη των προσπαθειών στον τομέα των νέων τεχνολογιών, καθώς έγινε πολλού λόγος, θα βοηθούσε να σπάσουν δημιουργικά και τα υπάρχοντα μονοπόλια μέσω του προγράμματος Horizon 2020 για μια ευρωπαϊκή Silicon Valley. Παρ' όλα αυτά το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη αρχίσει να περικόπτεται. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα έπρεπε να γίνει ή να γίνει από του διαδόχους σα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now our last... Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάνιεν, τελευταίος. Και ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, θέλω και εγώ να σας συγχαρώ για τη δουλειά σας. Να μην σας συγχαίρονται μόνο οι σοσιαλιστές. 20 χρόνια με εδώ στο Κοινοβούλιο. Και έχω περάσει και την περίοδο του Φανμίρτ και του Μόντι και τώρα βλέπω μετά τον ε, ε, παράξερο εκείνο Φαν Μίρτ και τον καθηγητή Μόντι, έναν ρεαλιστή και πραγματιστή αλμούνια. Ίσως θα πρέπει για την περίπτωση του Google να δούμε μήπως υπάρχει δυνατότητα να καταπολεμήσουμε και να προσπαθήσουμε να κατακαιρματίσουμε τον τομέα αυτόν, όπως έγινε στις ΗΠΑ πολύ παλιότερα στο τομέα του πετρελαίου και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Γιατί διαφορετικά όσο μπορέσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο του μονοπωλίου. Και επίσης, όταν διατυπώνει μία προσφυγή ένας εμπλεκόμενος, ε, πώς εξετάζει η Επιτροπή ε, το θέμα αυτό. Ασχολείται με την κάθε προσφυγή ή περιμένει να φτάσει και να κρυφτεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ξέρετε τι εννοώ. Επίσης για το Nürburgring, στην περίπτωση Nürburgring, ξέρετε ότι έφτασαν από πλευρά σας κάποιες ε, παρατηρήσεις για απάντηση στις ε, τοποθετήσεις των εμπλεκομένων. Τι νομίζετε λοιπόν ότι θα πρέπει για την Φόρμουλα 1 να κρίνει τελικά εάν θα διεξαχθεί εκεί πέρα το δικαστήριο, δεν πρέπει εσείς να τοποθετηθείτε ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Και η τελευταία ομάδα ερωτήσεων θα λάβει απαντήσεις σύντομες, θα έλεγα λακωνικές. Πρώτα απ' όλα, για τον κύριο Νίτερ Μάιρ. Εγώ είμαι υπέρ της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών ευρημάτων και νομίζω ότι των νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και νομίζω ότι η απόφαση του δικαστηρίου μας δίνει τα σχετικά μέσα. Άρα θέλω το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν τη συζήτηση για τον σχετικό κανονισμό, κάτι το οποίο θα εξασφαλίσει ιδεώδεις λύσεις και για τον ε, χρήστη και για τον ε, έμπορο. Ε, είπα ποιο είναι το κόστος 10 δις ευρώ το χρόνο από τις συνθήκες που επικρατούν τώρα στη σχέση με τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα ΜΥΦ. Εγώ αυτό δεν το βλέπω πουθενά στο λογαριασμό μου όταν πληρώνω. Δεν βλέπω δηλαδή πόσα μου χρεώνονται επειδή χρησιμοποιώ την κάρτα. Και επίσης στον τομέα αυτών με κάθε σεβασμό, ό,τι πρόκειται για, τις, ε, για το χώρο των πληρωμών, των τραπεζών κτλ. Από το 2007 και μετά νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει μια σειρά ισχυροτάτων, ε, έχουν αναπτυχθεί μάλλον μια σειρά ε, ισχυροτάτων επιχειρημάτων που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στον, στην αυτορύθμιση. Γι' αυτό και πρέπει να περάσουμε στον κανονισμό. Δεν είναι όλοι οι κανονισμοί η, η καλύτερη λύση πάντα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι. για τον κύριο Κόφωτ. Κρατικές ενισχύσεις και περιφερειακές ενισχύσεις. Τελευταίες ε, κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις πριν από ένα περίπου χρόνο ή φέτος ακόμη, δεν θυμάμαι πότε υιοθετήθηκαν, ίσως πέρσι. Στι τελευταίε αυτέ τι κατευθυντήρε γραμμέ, λοιπόν, είχαμε θεσπίσει πολύ συγκεκριμένε προποθέσει για να αποφύγουμε τι ε, επανεγκατεστάσει των ε, επιχειρήσεων που θα στηρίζονταν σε χρήμα από κρατικές ενισχύσεις. Δεν μπορούμε να συστήσουμε το θέμα της κρατικής ενίσχυσης υπό άλλη σκοπιά, αλλά αυτή η έννοια και βέβαια το θέμα των περιφερειακών ενισχύσεων που είχε αναλάβει ο αρμόδιος συνάδελφος μαζί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το είδαμε πολύ μεγάλη προσοχή και με τον Ιωάννης Χάν συνεργαστήκαμε πάρα πολύ προσεκτικά ώστε να αποφύγουμε τις ε, της, ε, τις ασυμβατότητες ε, σε σχέση με το θέμα των περιφερειακών ενισχύσεων και να αποφύγουμε τις καταχρήσεις έτσι. Για τον κύριο Σφάπ, σας ευχαριστώ θερμά για το ρόλο που είχατε στη συζήτηση της ιδιωτικής αποζημίωσης, ε, για όλη τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, για την Google. Και με κάθε σεβασμό πολιτικός είμαι και ξέρετε ότι ο πολιτικός με βάση την κοινή γνώμη αμείβεται. Ως εκ τούτου την σέβομαι την κοινή γνώμη. Αλλά δεν μπορώ στην κυρία Βεστάγκερ παρά να... Δεν μπορώ στην κυρία Βεστάγκερ να αφήσω σαν παρακαταθήκη μία πρόταση που θα λέει ας κρίνουμε τι θα κάνουμε με την Google ή κάποια άλλη μεγάλη και μονοπωλιακή θέση με βάση το τι θα πει η κοινή γνώμη. Όχι. Θα κοιτάξουμε την ομοθεσία, την κατάχρηση της πόσης θέσεως, τα επιχειρηματά μας, τον ανταγωνισμό και με βάση αυτά θα λάβουμε την απόφαση. Το άρθρο 7 ήταν η καλύτερη λύση. Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητάμε για χρόνια. Στην περίπτωση της Microsoft, που ερευνούσαμε επί 16-17 χρόνια εδώ και ακόμη πιο πριν στις ΗΠΑ, αξιοποιήθηκαν και τα δύο μέσα. Και του άρθρου 7 και δύο φορές παραβίασε του όρου του άρθρου 7 η Microsoft και καταδικάστηκε να πληρώσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ για το γεγονό ότι παραβίασε απόφαση του άρθρου 7 που της είχε επιβάλει 500 εκατομμύρια ευρώ. Άρα πλήρωσε το διπλάσιο σε πρόστιμο επειδή δεν σεβάστηκε η απόφαση του άρθρου 7 το 2009 με την Έλλη Κρούς. Επίτροπο. Και λήφθηκε η απόφαση του άρθρου 9 που πάλι παραβίασε και τότε της επέβαλα εγώ 560 εκατομμύρια ευρώ. Εν όλο δηλαδή κατέβαλε μεγαλύτερα πρόστιμα για παραβίαση ε, προηγουμένων αποφάσεων από ό,τι ήταν το αρχικό πρόστιμο. Αυτό για να σας πω ότι ο ανταγωνισμός δεν κρίνεται με ιδεολογία, αλλά με τρόπο ρεαλιστικό και πραγματιστικό. Και στον κύριο Ρωσάτη είπα, στην περίπτωση της Γκάσπρομ, είχαμε την ευκαιρία να διαρευνήσουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε απόφαση του άρθρου 9 Ανοίξαμε λοιπόν την πόρτα να κοιτάξουμε αυτή την επιχειρηματολογία, αλλά τώρα δουλεύουμε με το άρθρο 7, γιατί τη Motorola και τη Samsung, αποφάσεις που ελήφθησαν την ίδια ημέρα για ανάλογο τύπου παραβιάσεις, η απόφαση Samsung ήταν του 9, ενώ η απόφαση του, της Motorola ήταν επί βάση, του άρθρου 7. Ε, εν πάση περιπτώσει όμως να συζητάμε την ουσία και όχι τα μέσα περισσότερο και τις διαδικασίε. Για την υποστήριξη μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορώ να σας πω ότι με τα μέσα των κρατικών ενισχύσεων έχουμε τουλάχιστον τρία θετικά μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την οδηγία για τη χρηματοδότηση, κατευθυντήρες γραμμές για τη χρηματοδότηση κινδύνου, που σαφέστατα υποστηρίζει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω μη τραπεζικών συστημάτων χρηματοδότησης. Και αυτό νομίζω το απάντησα και νωρίτερα με τον κύριο ερώτηση του Φερνάντες. Έχουμε λοιπόν τι κατευθυντήριε γραμμέ, έχουμε τι περιφερειακέ κατευθυντήριε γραμμέ, που θα μπορούσαν να περιορίσουν ε, και ξέρω ότι για κάποιου βουλευτέ ε, οι περιφέρειε εκλογικέ ε, έχουν εκφραστεί αντιρρήσει ω προ τη διοχέτευση των κρατικών ενισχύσεων προ τι μεγαλύτερε επιχειρήσει. και έτσι όρισα εγώ όριο ανώτατο γιατί θεωρώ ότι οι περιφερειακέ ενισχύσει αυτέ θα πρέπει να στοχεύουν στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή νέων πρωτοβουλειών κτλ. Και μετά υπάρχει ο κανονισμό για τη γενική εξαίρεση προστασία ο οποίος θεσπίζει ένα πολύ πιο απλό τρόπο για την ανάλυση θεμάτων κρατικών ενισχύσεων, ακόμη και από το ίδιο το κράτος μέλος, χωρίς προειδοποίηση ή ε, εξάντε προειδοποίηση, ειδοποίηση, η εξαντε προειδοποιηση καλύτερα. Και αν θυμάμαι καλά, τα δύο τρίτα της κρατικής, των κρατικών ενισχύσεων που θα αναλυθούν θα εξαιρεθούν από την ε, από τη διαδικασία παρεμπόδιση. Ε, στη συνέχεια, αν υπάρξουν προσφυγές, θα το κοιτάξουμε προσεκτικά, αλλά σε πρώτη φάση επιτρέπουμε να ε, προχωρήσουν. Κατά τα άλλα, ναι, είμαι μεταρρυθμιστής, είμαι υπέρ των ε, ε μεταρρυθμίσεων, αλλά δεν πρέπει να γίνονται μεταρρυθμίσεις δεν και καλά. Θέλω να γίνονται όταν γίνονται μεταρρυθμίσεις για τον καλό σκοπό και όχι για τον κακό σκοπό, γιατί μερικές φορές γίνονται και για κακό σκοπό οι μεταρρυθμίσει. Και έχουμε παραδείγματα και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, στην κάθε χώρα ο καθένας μας τέτοιων περιπτώσεων. Ε, κύριε Λάγκεν, ευχαριστώ πολύ για τα ευγενή σας λόγια. Η απόφαση που αναφέρατε για την Urban Green ε, θα υιοθετηθεί την 1η Οκτωβρίου, άρα θα, την θα μπορέσετε να την αναλύσετε σε μερικές μέρες λεπτομερέστερα. Η δε κοινή γνώμη, η δε πρόταση για, την, ε, για τον κατακαιρματισμό της Google. Θα σας πω το εξή. Ναι, και είστε φίλος και Γερμανός. Γερμανός φίλος δηλαδή. Θα σας πω το εξής. Τη μέρα που θα μάθω ότι δέχονται την αποδεσμοποίηση οι σιδηρόδρομοι, οι εταιρείε ηλεκτρισμού, οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών και λοιποί φορείς, τότε μπορώ να συζητήσω και τον κατακαιρματισμό της Google, αλλά όχι πιο πριν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, τον Αντιπρόεδρο Αλμούνια και ολόκληρη την Επιτροπή βεβαίως. Ευχαριστούμε για όσα κάνατε όλα αυτά τα χρόνια στην Επιτροπή. And again for your excellent cooperation. Ευχαριστούμε και πάλι για την εξαιρετική συνεργασία με την Επιτροπή μας. Adios, now we start our session uh, και τώρα ξεκινάμε ε, το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Καταρχήν να καλωσορίσω όλους τους εκπρόσωπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια σε αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων Πολύ επίκαιρη ανταλλαγή απόψεων. Μέσα στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμένου για το 2014 που τώρα έχει φτάσει σε κρίσιμη φάση ε, δηλαδή είμαστε στην υιοθέτηση των ειδικών συστάσεων από το Συμβούλιο για την κάθε χώρα και την υιοθέτηση των εθνικών προϋπολογισμών από τα κράτη, μέλη. Uh, Έχουμε εμείς την έκθεσή μας συντάξει, την οποία και θα συζητήσουμε. Και στόχος αυτής της συνεδρίασης είναι ακριβώς να συνδεθεί η συζήτηση επί της έκθεσης ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες με μια συζήτηση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων ώστε να συγκεντρώσουμε τις συμβολές πριν να οριστοκοποιήσουμε την έκθεσή μας και συντάξουμε τη συμβιβαστική μας έκθεση. Να σας θυμίσω ότι δεδομένου το μεγάλο αριθμό μελών που είναι παρόντες και για να διευκολύνουμε ε, την συμμετοχή και την εκπροσώπηση όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων, μόνο ένας ανά Εθνικό Κοινοβούλιο θα πάρει το λόγο καταρχήν Εάν ωστόσο υπάρξει αρκετό χρόνος μετά από ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων παρατηρήσεων, τότε θα μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο και σε άλλον έναν από το ίδιο κοινοβούλιο. Έχουμε 21 γλώσσες σήμερα και χρησιμοποιείτε ε, τις ε, κάρτες ομιλίας για να διευκολυνθεί η συζήτηση. Εάν τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων ή το μέλη του ε- Ευρωκοινοβουλίου θέλουν να μιλήσουν, παρακαλώ συμπληρώστε την κάρτα ομιλίας και δώστε τη στους κλητήρες. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τιμπάκερ που είναι ο εισηγητής για να μας παρουσιάσει την εκθεσία του. Μάξιμουμ έχει 10 λεπτά στη διάθεσή του και μετά θα πάρουν το λόγο οι σκιώδεις εισηγητές και στη συνέχεια τα μέλη των Εθνικών και του Ευρωκοινοβουλίου. Κύριε Ντεμπάκερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και εγώ από το πλευρά μου θέλω να καλωσορίσω εδώ τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, τους εθνικούς βουλευτές. Είναι πάντοτε καλή ευκαιρία να, μπορούμε να συζητήσουμε την έκθεση που προετοιμάζει το Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις συγκεκριμένες συστάσεις μαζί σας με τα, εθνικά μέλη, τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων για να έχουμε τις απόψεις σας έτσι ώστε όταν εδώ εμείς ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες προσπαθούμε να βρούμε κάποια συμβιβαστική λύση, να μπορούμε να λάβουμε υπόψη και τους δικούς τους προβληματισμούς. Όπως είπε ο Πρόεδρος, η έκθεσή μας ε, είναι πολύ επίκαιρη γιατί ε, και στο Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο συνεχίζεται η διαδικασία υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το έχουμε αυτό βέβαια κάνει και στο παρελθόν. Οι εκθέσεις αυτές είναι πάντοτε πολύ σύντομε και επί της ουσίας ε, δεν έχουμε κανένα ένα ευχολόγιο, αλλά εστιάζουμε σε κάποια κρίσιμα θέματα που θεωρούμε σημαντικά αφού έχουμε λάβει υπόψη και τις δικές σας απόψεις. Εν συντομία θα σας παρουσιάσω την έκθεση που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Ξεκινάμε λέγοντας και περιγράφοντας μάλλον την οικονομική κατάσταση στην οποία εξακολουθούμε να βρισκόμαστε και σήμερα. Είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε κάποια πολύ ευάλωτη ε, εύθραυστη ε, πρόοδος, αλλά βέβαια ξέραμε πως ήταν πολύ δύσκολο να συντηρηθεί και γι' αυτό και τους τελευταίους μήνες είδαμε ότι όντως δεν ήταν βιώσιμη, δεν στηρίχθηκε και είμαστε σε πολύ επικίνδυνα νερά πάλι. Αυτό ε, αναφέρεται στην εισαγωγή, στην έκθεση και εδώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο επισφαλής είναι η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα αργή ανάπτυξη και τεράστια ανεργία σε πολλές χώρες. Όπως είπα η έκθεσή μου βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Η οικονομική διακυβέρνηση και το πλαίσιό της ωστόσο θα πρέπει να διατηρηθούν ναι, εφόσον είμαστε ακόμα στα μέσα της κρίσης και χτες μάλιστα μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον κύριο Ντράγκη που μας είπε ότι θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο το να αλλάξουμε τώρα το οικονομικό πλαίσιο και το πλαίσιο διακυβέρνησης γιατί έτσι δώσαμε κάποιες κατευθύνσεις στην αγορά. Θα ήταν λάθος λοιπόν ε, να αλλάξουμε κάτι σε όλα αυτά. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τη μέγιστη ευελιξία που δίνεται στο πλαίσιο της ε, διακυβέρνησης ε, ε, και Φυσικά υπάρχει και αιρεσιμότητα στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν οι όροι, οι προϋποθέσεις. Θα πρέπει να ε, εστιάσουμε στην εφαρμογή των διαστατικών μεταρρυθμίσεων, η οποία είναι πολύ σημαντική και φυσικά στο τέλος μιλάμε και για την ευφυή δημοσιονομική εξυγίανση. Ε, τα κράτη μέλη ήδη κάνει μεγάλες προσπάθειες και θα πρέπει κάπως να μπορέσουμε να τις ελαφρύνουμε από αυτές, αυτό τα βάρη. Επόμενος προβληματισμός είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί στα κρατη για να εφαρμοστούν οι διαρθωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει όμως και η πτυχή της νομισματικής πολιτικής, η οποία ωστόσο από μόνη της δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Και ο ίδιος ο κύριο Ντράγκη είπε ότι μπορεί ακόμα περισσότερο να προχωρήσει σε προσπάθειες, ωστόσο μόνη της ε, η νομισματική πολιτική δεν θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση στην κρίση έξοδο από την κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τα αριθμιστικά πλαίσια που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίσουμε πως και εκεί ε, ας πούμε για τις τράπεζες, τις δημοσιονομικές, τις χρηματοπιστωτικές αγορές να υπάρχουν αρκετές δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν τα μέσα που προσφέρει η ΕΚΤ ώστε να εξέλθουν από την κρίση. Τρίτη μου είναι αυτή η παρατήρηση στην έκθεσή μου. Ε, εστιάζουμε την προσοχή στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. Ε, χειρισμός και αντιμετώπιση του, δημοσίου, του ιδιωτικού μάλλον χρέους δεν μιλάμε μόνο για δημόσιο χρέο, αλλά και για ιδιωτικό χρέο σε αύξηση των ε, δυνατοτήτων χρηματοδότηση και τονίζουμε τι καινοτομίε που θα πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε μόνο νέα σχήματα, νέε ιδέε, νέε επιχειρήσει, αλλά ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να κατακτήσουν την αγορά και θα σημάνουν τη διαφορά στις ζωές των συμπολιτών μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και πάλι να επιστρέψουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή ενέργεια, κλίμα, ψηφιακή ατζέντα και ούτω καθεξής. Τελευταία μου παρατήρηση εστιάζει στη πολύ σημαντική υπόθεση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και δημοκρατικού Γι' αυτό ευρίσκεστε και εδώ, ώστε να είμαστε βέβαιοι πως η συζήτηση αυτή θα γίνει όσο γίνεται πιο δημοκρατικά. Αναφέρομαι την έκθεση της Τρόικα, ε, για την Τρόικα που συνετάχθη από το Κοινοβούλιο και επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η Τρόικα στο παρελθόν και επίσης θυμίζει το γεγονός ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα στο πλαίσιο της κοινοτικής μεθόδου και μέσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο αναφέρουμε και το γεγονός ότι η Ευρωζώνη θα έπρεπε να αντιπροσωπεύεται και να εκπροσωπείται μάλλον σε διεθνείς οργανισμούς ώστε να έχει καλύτερο και μεγαλύτερο αντίκτυπο εκεί. Έμφαση δίνεται λοιπόν στο πλαίσιο διακυβέρνησης που έχει δημιουργηθεί, στη χρήση της μέγιστης ευελιξίας τα κράτη-μέλη να ιδιοποιηθούν τις συστάσεις του Συμβουλίου και να τις εγκρίνουν τις συστάσεις αυτές τις ίδιες ανά χώρα στο Συμβούλιο γιατί δεν έχει νόημα δύο μέρες μετά να λένε άλλα λόγια στις πρωτεύουσε. Πρόκειται για συστάσεις τις οποίες συντάσσει η Κομισιόν αλλά τις εγκρίνει το Συμβούλιο και άρα όλα τα κράτη-μέλη και άρα θα πρέπει να σημαίνει ότι συμφωνούν και εφαρμόζουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτά αυτή τη στιγμή έχουν μείνει πίσω, μόνο το 10 με 15% των συστάσεων έχουν εφαρμοστεί και ε, δεν, ε, για το 40-45% δεν έχει καν ξεκινήσει η σχετική συζήτηση. Οπότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει περισσότερο να ιδιοποιηθούν, όπω είπαμε, αυτέ τι συστάσει και να τι θέσουν σε εφαρμογή. Προσβλέπω λοιπόν στη συζήτηση και στη συμβολή σα και είμαι βέβαιο ότι τα μέλη των, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν ασχοληθεί με τη σύνταξη εκθέσεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα λάβουμε υπόψη όλε τι συμβολέ σα όταν θα συζητάμε την τελική εκδοχή τη εκθεσή μα τι επόμενε εβδομάδε και θα είμαστε, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στι συμβαστικές ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες. Σα ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή και δίνω το λόγο στους κοιόδη των πολιτικών ομάδων. Πρώτος είναι ο κύριος Ντάριο Ροζάτη. Και σας υπενθυμίζω ότι έχετε το πολύ τρία λεπτά για την κάθε παρέμβαση. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Και επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή κύριο Ντεβάκα Για την έκθεση το ΕΛΚ ως ομάδα συμμερίζεται προς από τις σημαντικές ε, παρατηρήσεις της εκθέσεως και νομίζω ότι τίνει προς την ορθή κατεύθυνση έτσι ώστε να έχουμε εν τέλει μια έκθεση η οποία θα καλύπτει τα πιο σημαντικά ζητήματα. Εδώ έχουμε μια από τις πρώτες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και είναι πολύ σημαντικό εδώ να υπογραμμίσουμε πως οι συστάσεις για την κάθε χώρα θα πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη σοβαρά από τα κράτη-μέλη. Εδώ πέρα λοιπόν αυτή η έννοια του ownership, δηλαδή να ενστερνίζονται ε, τις συστάσεις οι χώρες που τις αφορούν, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει δηλαδή να τις ε, μεταχειρίζονται σαν προγράμματα δράσης δικά τους. Και αυτό νομίζω ότι μπορούν να το ε, μεταφέρουμε και προς τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων, δηλαδή να τους ζητήσουμε καταρχάς να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις συστάσεις αναχώρα και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται πολύ περισσότερο στη διαδικασία αυτή. Ίσως λοιπόν μπορούμε να ε, προβλέψουμε μια διαδικασία συμμετοχής και των Εθνικών Κοινοβουλίων σε κάποιο στάδιο ώστε να είναι ενήμερα τα εθνικά κοινοβούλια, τι είδου συστάσει αναχώρα προετοιμάζει το κοινοβούλιο και όταν το Συμβούλιο είναι έτοιμο να λάβει τελική απόφαση, θα είναι και τα εθνικά κοινοβούλια πιο εξοικειωμένα με τι συστάσει, με τι προτάσει. Ένα άλλο θέμα βεβαίω είναι ότι δεν μπορεί η νομισματική πολιτική μόνη της να δώσει τις λύσεις, θα πρέπει να υποστηριχθεί και να συνοδευτεί και από μια ε, δημοσιονομική, μια ε, φορολογική πολιτική κατάλληλη και το κατάλληλο μείγμα πολιτικής. Για να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Όλα αυτά έχουν συζητηθεί κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μας με τους λοιπούς και οδησηγητές. Είμαστε στη φάση της προετοιμασίας τελικής εκθέσεως, η οποία εκτιμώ θα βοηθήσει και τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο να συντονίσουν ακόμη περισσότερο την πολιτική τους. Καλώς, σοσιαλιστές, δημοκράτες, τι Σάνε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και εγώ από πλευρά μου τον κύριο Ντεμπάκερ για τη δουλειά του. Βλέπω ότι έχει λάβει τη σωστή ε, κατεύθυνση η έκθεση. Τόσο εγώ όσο και άλλοι συνάδελφοι τη ομάδα μου έχουμε καταθέσει τροπολογίες όπως είχαμε υποσχεθεί. Οι συμβαστικέ λύσει που διαγράφονται νομίζω είναι πολλά υποσχόμενε Και στις περισσότερε περιπτώσει καλύπτουν τις ε, προσδοκίες των σοσιαλιστών δημοκρατών ήδη σε αυτό το στάδιο. Αντί λοιπόν να τοποθετηθώ σε σχέση με το πρώτο ε, σκαρίφημα της εκθέσεως, θα ήθελα να δώσω κάποιες γενικές κατευθύνσεις που πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση, θα πρέπει να τροποποιηθούν μέσα στην έκθεση. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι οι περιορισμοί θα μπορούσαν να φέρουν ε, την ε, ανάκαμψη στην Ευρώπη από μόνοι τους. Οι περιορισμοί οι ίδιοι, η λιτότητα δηλαδή, έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν φέρνει λύσεις. Υπάρχουν δε κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες ε, βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στις κοινωνίες μας. Δεν πιστεύουμε λοιπόν πως είναι σωστό να αποδίδεται υπερβολικά μεγάλο ρόλο στην έκθεση για το ζήτημα, στο ζήτημα της ιδιωτική ε, περιουσίας. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε τώρα για την κρατική περιουσία. Είναι αυτό το αντικείμενο στην ανάλυση της εκθέσεως. Από την άλλη με χαρά σημειώνουμε ότι σε αυτό το σημείο όπως και σε άλλα έχουμε επιτύχει ε, συμβαστικές λύσεις ή τίνουμε προς συμβαστικές λύσεις που θα είναι ικανοποιητικές για τους πάντες. Υπάρχουν βέβαια κάποια αισθήματα εκκρεμή που μπορούν ωστόσο την Πέμπτη με τη συνεδρία των συντονιστών να επιληθούν. Και πάντως είμαι αισιόδοξο γιατί βλέπω ότι είναι πολύ υποσχομένο το πνεύμα με στο οποίο δεξάγονται αυτές οι συνομιλίες. Θα ήθελα να επισημάνω τώρα την περιγραφή της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας που για μας αποτελεί ε, κύρια προτεραιότητα, κέρια προτεραιότητα. είναι γνωστό ότι έχουμε εξασφαλίσει την κατάθεση μιας συμβαστικής τροπολογίας που πιστεύουμε μπορεί να εγκριθεί. Ε, θέλω να, να ευχαριστήσω τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων για την εμπλοκή τους σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και τις δικές τους θέσεις για τις συστάσεις αναχώρα και το εξάμεινο γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από το ΙΣΙΑ, σαν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπα στην πρώτη συζήτηση, έχει κάνει καλή δουλειά ο κύριος Δεμπάκερ, αναφέρει τα βασικά σημεία που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και έχει κάνει και παρατηρήσεις πολύ σωστές και εύστοχες για το πού θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εξυγχρονισμού. Παράδειγμα, στη χώρα μου, τη Φιλανδία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση και σε ε, ε, άλλα συστήματα χρειάζεται πηγόντως μεταρρύθμιση. Και επίσης ε, εξετάζει και τις αλληλεπιδράσεις των μεταρρυθμίσεων. Συμφωνώ γενικότερα με τον εισηγητή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τις οικονομίες του στα κράτη-μέλη. Και συμφωνώ κατά κύριο λόγο με τις λύσεις που προτείνει. Εκεί που διαφωνώ ε, σε κάποιο βαθμό είναι ο ρόλος που θα πρέπει να κληθεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λυθούν τα προβλήματα. Ε, για τους συμβιβασμούς, οι συμβαστικές τροπολογίες ε, παραμένουν ορισμένες από εμά απαράδεκτες και S και V για τους συντηρητικούς. Είμαστε κατά όλων των συμβιβασμών που φιλοδοξούν να κάνουν τις συστάσεις αναχώρα πιο δεσμευτικές προς τα κράτη-μέλη μεταξύ αυτών είναι για παράδειγμα και η ιδέα ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους δεν συμμορφώνονται προς τις συστάσεις αναχώρα. Οι συστάσεις αναχώρα είναι, όπως ξεκάθαρα τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συστάσεις που βασίζονται σε λεπτομερή ανάλυση της κατάστασης σε κάθε χώρα και δίνουν μια καθοδήγηση κατεύθυνση και το τονίζω αυτό για το πώς ε, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Συστάσεις είναι και ως τέτοιες θα πρέπει να τις ε, εξετάζουμε και να τις μεταχειριζόμαστε και δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να τιμωρούνται επειδή δεν τις ακολουθούν. Με άλλα λόγια, στη δημοκρατία η οικονομική πολιτική θα πρέπει να αποφασίζεται από πολιτικούς οι οποίοι εκλέγονται από λαούς δεν μπορούμε να δώσουμε, να χωρίσουμε και άλλες εξουσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν είναι εκλεγμένη για να ελέγχει, να έρχεται και να τιμωρήσει εκλεγμένους πολιτικούς που ασκούν πολιτική στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. E. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρίζα Ματίας από την ΚΟΕ. E. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του που είναι υποδειγματική. Αυτό δεν είναι καινούριο. Έχουμε διαφορετικές απόψεις ε, ε, βέβαια για το πώς αναλύουμε αυτή την υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, όχι μόνο στο τι γίνεται αλλά και στις προτάσεις που γίνονται. Ο εισηγητής Θεωρεί ω προπόθεση πω οι χώρε που εφάρμοσαν τι μεταρρυθμίσει, τι διαρθρωτικέ, είχαν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τι οικονομίε του όσον αφορά την ανάπτυξη, την ενίσχυση της σε της δημοσιονομικής. Εμείς διαφωνούμε κάθετα, απόλυτα, δεν είναι αλήθεια. Οι χώρες οι οποίες προέβησαν στις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις ε, βρίσκουν την οικονομία τους τελείως κατεστραμμένη. Έχουν σχεδόν μηδενική ανάπτυξη, μηδενική... Ε, ο, ο, προϋπολογισμός τους έχει καταβαραθρωθεί ε, και... όπως καταλαβαίνετε αντίθετα με τα όσα λέει η έκθεση δεν νομίζω πως μπορούμε να μιλήσουμε για οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο γιατί η λιτότητα απέτυχε και η λιτότητα η οικονομική ε, επιδίνωσαν τα προβλήματα της οικονομίας, της εθνικής οικονομίας της κάθε χώρας που ποτίθεται ότι θα τα έλυναν. Και βάθυναν ακόμη περισσότερο την ύφεση. Δεν έχουμε λοιπόν περιθώριο ελιγμού, δημοσιονομικού ελιγμού και ακόμα και στις οικονομίες που εφαρμόστηκαν οι συστάσεις δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης. Αντίθετα από αυτά που προτείνει ο εισηγητής λοιπόν, πιστεύουμε πως ε, ε, μόνη περίπτωση για να είναι βιώσιμες βιώσιμος εθνικός προπολογισμό είναι να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να υπάρξει ανάπτυξη. Αλλά κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται με βάση τα όσα προτείνονται. Συνεχίζεται η ίδια πολιτική και είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει στην συντήρηση των προβλημάτων που υπάρχουν τώρα. Οι προτάσεις λοιπόν που υποβάλλονται εξακολουθούν να επικεντρώνονται στις δαπάνες και στην απορρίθμιση του, της εργασιακής αγοράς και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι σε ύφεση με πολύ αδύναμη ανάπτυξη, αλλά κάθε φορά που υπάρχει έστω και μια μικρή ανάπτυξη, μια μικρή ανάπτυξη, ε, δεν οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια ριζική αλλαγή των ε, προσανατολισμών. Πράγμα που δείχνει ότι είναι σημαντικό οι συγκεκριμένες συστάσεις που γίνονται στις χώρες να δίνουν όλο ένα και μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτικές στον τομέα της ζήτησης. Δηλαδή για να ενισχυθεί ο τομέας της ζήτησης δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής και πολιτικές που να οδηγούν στην αύξηση των μισθών. Η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας και η επισφάλεια στην απασχόληση δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα, ούτε πρόκειται να οδηγήσει σε βελτίωση της οικονομίας. Οι θέσεις μας είναι λοιπόν αντίθετες και τελευταία να ότι υπάρχει και το πρόβλημα, το βαθύ πρόβλημα το δημοκρατικό. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αφαιρεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια δυνατότητα, τη δυνατότητα να αποφασίζουν για πολιτικές τόσο θεμελιώδεις όπως είναι η δημοσιονομική πολιτική της κάθε χώρας. Ευχαριστώ τον εισηγητή όπως είπα για τον εισηγητή, αλλά δεν είναι δυνατόν να βρούμε συμβιβαστική λύση εδώ. Ευχαριστώ. Από τους πράσινους ο Μπάς Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω η συζήτηση αυτή δείχνει στους εθνικούς βουλευτές συναδέλφους μας πόσο δύσκολο είναι να πετύχεις πλειοψηφία ε, ο, ο εισηγητής λέει εύκολο είναι. Ναι, για να δούμε. Βλέπετε ότι υπάρχουν δύο διαχωριστικές γραμμές πάνω κάτω για αυτή την έκθεση. Ε, μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει αριστερή πτέρυγα του Κοινοβουλίου που είναι πολύ επικριτική για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η οικονομική διακυβέρνηση. Και μέχρι τώρα βασικός μας στόχος ήταν να μειωθεί το εργατικό κόστος και να συμπιεστεί και να δούμε μόνο το δημόσιο χρέος ενώ όλοι αναγνωρίζουν βεβαίως ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το ιδιωτικό χρέος και χρειάζεται πιο ισορροπημένη προσέγγιση και όταν ε, ε, κεντρώνεσαι στη συμπίεση του εργατικού κόστους δεν είναι κοινωνική η προσέγγιση αυτό που κάνει τώρα η Ευρώπη και ε, εστιάζεται στη λιτότητα. Ελπίζω σιγά σιγά μια πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι δεν είναι λύση. Αλλά πρέπει να βρούμε μια πλειοψηφία. Υπάρχει αυτή η διαχωριστική γραμμή δεξιά-αριστερά. Η άλλη είναι η σημασία. Πόσο σημαντική θεωρείς δηλαδή την οικονομική διακυβέρνηση και αν θέλεις περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές και καθοδήγηση όχι. Και ο συνάδελφός μου από τη Φιλανδία, ο γνήσιο φιλανδό πρώην και νυν πραγματικός Φιλανδός, δεν ξέρω τι στο καλό Φιλανδός είναι πια, ε, Είπατε ότι ωραίο το ευρώ και η Ευρώπη και καλό να το έχουμε, αλλά να μην χρειάζεται κανένα συντονισμό. Άρα μήπως δεν θέλετε καθόλου το ευρώ να το πείτε. Ορισμένοι στην ομάδα σας το θεωρούν, αλλά το λένε. Και ε, εκεί υπάρχει άλλη μια διαχωριστική γραμμή. Υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της... Ε, οικονομικής διακυβέρνησης και το είπε και ο εισηγητής, αλλά για να το πετύχει αυτό χρειάζεται και λίγους αριστερούς. Και τώρα βρισκόμαστε στα μέσα των διαπραγματεύσεων για να γίνει η έκθεση πιο ισορροπημένη ο Φιλίπ, τι να κάνει ο άνθρωπος, ο καημένος φιλελεύθερος είναι ε, και από, από γεννησιμιού της η έκθεση έχει αυτή τη φιλελεύθερη κοπή και λέει ότι είναι εντάξει ε, η οικονομία και βρισκόμαστε στην ανάκαμψη. Ναι, αλλά στις διαπραγματεύσεις του είπαμε μην είσαι τόσο υπεραισιόδοξος δεδομένων και των πιο πρόσφατων εξελίξεων. Χρειάζεται μια αναπροσαρμογή αυτό και επίσης η μεγάλη λύση δεν πρόκειται να έρθει από τις ιδιωτικές επενθύσεις. Γνωρίζουμε όλοι ε, τι γίνεται η μείωση των επενδύσεων είναι και από την κρατική πλευρά και από την ιδιωτική. Καλά, τώρα δεν θα μπούμε στη γενική συζήτηση ποιε είναι οι καλύτερε επενδύσει ιδιωτικέ ή και τι δύο χρειαζόμαστε και θα πρέπει και αυτά να τα λέει πιο ισορροπημένα η έκθεση. Ε, Πάντω καλά πάνε οι διαπραγματεύσει και αφού χρειάζεται αυτή την πλειοψηφία υπέρ της οικονομικής διακυβέρνησης, χρειάζεται και την αριστερά, οπότε μετράει και αυτό στα κουκιά. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο. Η σημερινή κατάσταση και το πρόβλημα ποιο είναι. Μέχρι τώρα ουσιαστικά επικεντρωθήκανε στο, στη συμπίεση και τη μείωση του εργατικού κόστους. Αλλά χρειάζεται μια ισορροπία. Αλλά πρέπει να δούμε και το κόστος του κεφαλαίου. Πώς χρησιμοποιούμε τους πόρους με αποδοτικό τρόπο και με οικονομία. Συμπέρασμα, Πρόεδρε. Αυτό που θέλουμε όλοι στο τέλος είναι περισσότερες ε, και ειδικότερες συστάσεις αναχώρα για τη φοροδιαφυγή. Άλλη μεγάλη πληγή όταν συζητούμε την οικονομική διακυβέρνηση και βλέπω εδώ μέσα μερικούς Ολλανδούς συναδέλφους Μήπως έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε με την Ολλανδία και με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και χαίρομαι που το έχουν υπόψη τους οι Ολλανδοί αυτό, συνάδελφοι τουλάχιστον. Ευχαριστώ Μπάς. Από την ομάδα EFTD, δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει, Σκιώδης είναι. Έχω ένα όνομα για να ολοκληρώσουμε το γύρο των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ευχαριστώ. Έχω ένα-δύο προβληματάκια με το κείμενο που ήδη όμως αναφέρθηκαν που λέει ότι έχει αρχίσει η ανάκαμψη ενώ σαφώς δεν έχει αρχίσει τίποτα τέτοιο. Ε, και άλλο ένα σημείο είναι ότι ζητά τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν την ε, ατζέντα μεταρρυθμίσεων την οποία υπαγορεύει, υπαγορεύουν τα ευρωπαϊκά όργανα ενώ είναι υπόλογα στις, ε, στο κοινοβούλιο, και στο, στο κοινοβούλιο τους οι κυβερνήσεις. Όλα αυτά υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ε, ένα νόμισμα ε, χρειάζεται μια κυβέρνηση και μια χώρα για να είναι συνεπής. Γι' αυτό και η Ευρωζώνη ε, είναι, στην Ευρωζώνη επικρατεί χάος αυτή τη στιγμή οικονομική συνοχή για να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ανάπτυξης. Δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμότητα ε, γιατί οι, οι λαοί θεωρούν ότι η εθνικότητά τους είναι η ταυτότητά τους. Ε, ο δρόμος έξω από όλη αυτή την κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Το ευρώ θα πρέπει να διαλυθεί. Ε, και θα πρέπει να προστατευτούν τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας στις αδύναμες πλευρές ε, περιοχές της χώρας. Η αποσύνθεση του ευρώ δεν θα είναι εύκολη, αλλά μέχρι ότου να γίνει κάτι, ε, ε, μέχρι να γίνει μάλλον δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Εγώ βέβαια είμαι σε προνομιακή θέση, γιατί είμαι εκτός της ευρωζώνης, αλλά εν πάση περιπτώσει διαφορετικά δεν θα διορθωθούν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ και αρχίσουμε τώρα με τις παρεμβάσεις και από τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα δώσω το λόγο σε δύο συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και δύο συναδέλφους από το Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτος ομιλητής είναι ο Χούμπερτ Φούξ από το Εθνικό Κοινοβούλιο της Αυστρίας. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων που προσκάλεσε τι αντίστοιχε επιτροπέ των Εθνικών Κοινοβουλίων για τη σημερινή συζήτηση. Περαιτέρω βήματα για την υιοθέτηση των διαδικασιών στον, ε, στη διαδικασία του, Ευρωπαϊ, του Αυστριακού ε, Προπολογισμού για την Αυστρία ειδικά θα χρειαστούν ε, περαιτέρω προσαρμογέ. Έχουμε κάνει μια αξιολόγηση τη πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση του προπολογισμού με την παρουσία προτάσεων για την εναρμόνιση των εθνικών δημοσιονομικών διαδικασιών προς τις ε, προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πράγμα το οποίο θα σημάνει ίσως, μπορεί να σημάνει ίσως και την ε, εντονότερη παρέμβαση και συμμετοχή στη δικασία του Εξαμήνου του Εθνικού Κοινοβουλίου κατά την προετοιμασία του προσχεδίου και την έκρηση του υπολογισμού, ε, αλλά και την εμπλοκή κατά την συζήτηση και υιοθέτηση, αλλά και κατά την υλοποίηση των συστάσεων. Η Επιτροπή των Προπολογισμών έχει ζητήσει από την αντίστοιχη υπηρεσία του Κοινοβουλίου να σχολιάσει ιδιαίτερα τις προϋποθέσεις για το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν κάποια μέσα για πιο έντονη εμπλοκή, όπως σε παραδείγματι η δυνατότητα να προσκληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει την αξιολόγηση του προσχεδίου του προπολογισμού, λύση που θα μπορούσε να αξιολογηθεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο επόμενος ομιλητής, η ομιλήτρια, είναι η Κάταλεν Σχόμπο από την Εθνική, από την Εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντική για μας αυτή η συνεδρίαση. στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που έχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα για το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Η στρατηγική 2020 και η υλοποίησή της έχουν συζητηθεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης της Ουγγαρίας. Πέρυσι, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν η πρώτη φορά που έγινε μια πρώτη αξιολόγηση για κάθε χώρα μέλος με, με τη συνέχεια που δόθηκε με τις συστάσεις αναχώρα που καταγράφουν το πώς τα πάνε και τι πρέπει να κάνουν ακόμα οι χώρες. Εμείς συζητήσαμε τις συστάσεις αυτές και οι σχετικές με την Ουγγαρία χρόνο με χρόνο βλέπουμε ότι επανέρχονται. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να υλοποιηθούν. Η κυβέρνηση μπορεί να συμφωνεί με τις ε, συστάσεις με κάποιες από τις συστάσεις, αλλά δεν συμφωνεί με όλες ε, στο θέμα της φορολογίας η παραδείγματη, η οποία είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαφοροποιείται σε αυτό από τις θέσεις του Γκρικού Κοινοβουλίου. Εφέτος όμως φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία ως, ως προς το πρόγραμμα δημοσίων έργων που χρειάζεται η Ουγγαρία. Και θέλω επίσης να σημειώσω ότι έχει η Επιτροπή δεχθεί πως έχουν βελτιωθεί, η Επιτροπή δέχθηκε πως έχουν βελτιωθεί συνθήκες απασχολησιμότητας των γυναικών. Ότι δηλαδή οι γυναίκες μετά τον το κετό και την άδεια ξαναεπιστρέφουν, έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη θέση εργασία τους. Η ανάπτυξη επίσης έχει αρχίσει να διαφαίνεται τους τελευταίους μήνες και Σημειώνουμε με ικανοποίηση την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ένα άλλο σημαντικό για μας θέμα είναι αυτό της ενεργού συμμετοχής των κρατών μελών στη δικασία. Έχουμε αποκλειστικό, ε, αποκλειστική αρμοδιότητα της έγκρισης του Εθνικού Προϋπολογισμού. Αυτό θέλω να υπογραμμίσω και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα δικά του μέλη και την Ιβάνα Μάλεντιτς Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων, όπως και τους ε, συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις ε, συστάσεις αναχώρα τις έχουμε συστήσει για πολύ καιρό και ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν. Εδώ λοιπόν έχει μεγάλη σημασία το τι στάση και θέση θα τηρήσουν τα εθνικά κοινοβούλια. Γι' αυτό και διαρωτώ με γιατί την υλοποίηση των εθνικών των συστάσεων αναχώρα την επιβλέπει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή στην ε, διαδικασία αυτή επαλήθευση τη υλοποίηση των Εθνικών Κοινοβουλίων, αφού οι Εθνικέ Αρχέ είναι αυτέ οι οποίε θα πρέπει να υλοποιήσουν τι συστάσει χώρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαίρετη έκθεση, αλλά και την κυρία Ντανούτα Χιούπνερ, η οποία με τι ε, τροπολογίε τη τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της διασύνδεσης της οικονομικής με την πολιτική ανάπτυξη, ε, συνοχής και ιδιαίτερα τονίζει το ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα διορθωτικά κονδύλια για την ενίσχυση των ε, οικονομικών πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων που ε, καταγράφονται με τις συστάσεις αναχώρα. Έτσι μπορεί η πολιτική της συνοχής να στοχεύσει πιο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε για την προσεχή περίοδο 2014-2020. Και εν τέλει, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εξή για μένα. Τα κύρια συστατικά της ανάπτυξης είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική εξυγένση και οι επενδύσεις. Αυτό όμως που συχνά συμβαίνει στα κράτη είναι ότι η δημοσιονομική εξυγίανση οδηγεί σε μείωση των ε, κινήτρων που δίνονταν για επενδύσεις και ως εκ τούτου μετριάζει σημαντικά τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων. Εγώ πιστεύω ότι τα κράτη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν επαρκή ευελιξία ώστε να αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα υλοποιήσουν τα σχέδια που έχουν ε, καταρτήσει και εφόσον αποδεικνύουν ότι τα ε, και όσο τα αποδεικνύουν βεβαίως ότι τα εφαρμόζουν αποτελεσματικά. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα περιθώριο για δημοσιονομική εξυγίανση μεγαλύτερο για τα κράτη και τις κυβερνήσεις, να μην πιέζονται ε, κατά τρόπον ώστε να λαμβάνουν μέτρα τα οποία παρεμποδίζουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και, την, ε, και τις επενδύσεις για την ανάπτυξη. Κυρία Φερέιρα, έχει το λόγο. Θα τα πω αγγλικά για να τα πω πιο γρήγορα. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για τη ε, δουλειά του. Καλωσορίζω τα Εθνικά Κοινοβούλια, διότι πιστεύω ότι αυτό που συζητούμε είναι μείζον θέμα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σημαίνει σημαντική αύξηση ε, της ισχύς και της εξουσίας διείσδυσης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στα σχέδια προϋπολογισμών και τους ίδιους τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας τι σημαίνει αυτό και ποιες οι συνέπειες των όσων αποφασίζουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση αυτή καθ' αυτή υπάρχουν στοιχεία που είναι θετικά όπως η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, η στρατηγική 2020, η κυλοποίησή της, αλλά το συμπέρασμα και η κεντρική ιδέα για μας, για την πολιτική μας ομάδα, θα εξαρτηθεί από το μήνυμα που θα δοθεί. Θα επιβεβαιώσει τη στρατηγική που ακολουθήθηκε ή θα συμπεριλάβει την ανάγκη αλλαγής και αναπροσαρμογής αυτής της πολιτικής. Τα πάντα λοιπόν θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των συμβαστικών διαπραγματεύσεων. Εμείς για παράδειγμα πιστεύουμε ότι εάν το τελικό αποτέλεσμα καταλήγει στη συνέχιση της ε, ε, ατζέντα και κυριαρχήσει η ανάκαμψη για μας δεν είναι εύστοχο η Ευρωζώνη αναπτύσσεται με ρυθμούς 0,8%, υπάρχει κίνδυνος αποπληθωρισμού και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες της αγοράς ε, δεν επιτρέπουν αυτή την ε, συνήθη ε, οικονομική, νομισματική μάλλον πολιτική και σκέφτονται έκτακτα μέτρα. Και η ανάκαμψη χρησιμοποιείται γενικά και αόριστα για τα πάντα. τελικά είναι πολύ περιοριστική η φεσιακή ατζέντα αυτή, πολύ γρήγορη, πολύ σκληρή και ε, έχει οδηγήσει σε αυτή τη στασιμότητα στην οικονομία ε, χωρίς καμία ζήτηση, με πολλές ανισορροπίες. Δεν υπάρχει ζήτηση ούτε για επενδύσεις ούτε για κατανάλωση. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει με κάποιο τρόπο. Και επίσης θα πρέπει να συμμορφώνονται οι χώρες με τις συστάσεις, αλλά τι σημαίνει αυτό. Για να συμμορφωθούν θα πρέπει να δούμε τι ποιότητα είναι αυτές οι συστάσεις και να έχουν συζητηθεί αυτά τα θέματα σωστά και σε βάθος. Εμείς έχουμε μεγάλες δυσκολίες να δεχτούμε προτάσεις τύπου δημόσιες επενδύσεις δεν είναι θετικές ενώ είναι ιδιωτικές. Τι έχουμε δηλαδή, καλές και κακές επενδύσεις, καλά και κακά έχουν και οι δύο, το έδειξε και η κρίση. Η ιδιωτική επένδυση δεν ήταν πάντα ο καλύτερος τρόπος. Ε, και υπήρχε και μεγάλος ήταν προσανατολισμένη στο μεγάλο κίνδυνο δηλαδή. Και δεν είναι λύση για την ευρωπαϊκή αγορά σε ένα παγκόσμιο κόσμο οι επενδύσεις που είναι σχεδόν μηδενικές. Ε, λοιπόν, θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά και να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις του εισηγητή με τους σκιώδεις μέχρι την τελική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ όμως για την ευκαιρία που έχουμε να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ Ελίζα. Και τώρα πάμε πάλι στα Εθνικά Κοινοβούλια. Μπιρούτε Βεσάιτε από τη Βολή της Λιθουανίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή και για τις συστάσεις σαν χώρα. Έχω να πω το εξής. Η Λιθουανία είναι από τις 10 χώρες με τις καλύτερες, μάλλον με τις χειρότερες επιδόσεις. Ε, στο παρελθόν και τώρα έχει αρχίσει να ανακάμπτει. Αν ρωτήσετε όμως τους Λιθουανούς αν τους αρέσει να ζουν στη Λιθουανία, οι περισσότεροι θα σας πούν όχι. Ε, θέλω να επιστήσω την προσοχή ε, του ε, εισηγητού ε, στις ανισότητες που αυξάνονται στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών είναι το μεγαλύτερο και ευρύτερο από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και Και επίσης υπάρχει και το πρόβλημα αύξησης της ε, ε, φτώχειας μεταξύ των εργαζομένων. Έχουμε εργαζομένους φτωχούς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το κοιτάξει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εισηγητής. Ε, έρχομαι τώρα στο φορολογικό και στη φοροαποφυγή και στη φοροδιαφυγή. Υπάρχει ένας φόβος να φυγούν αυτά και να μεταρρυθμιστούν τα συστήματα. Αν θέλουμε ένα δημοκρατικό καθεστώς, εάν δεν θέλουμε να ανεβαίνει η ακροδεξιά και οι λαϊκιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες μεταρρυθμίσεις που αναγκαστικά μετατίθενται στο μέλλον λόγω της Ουκρανορωσικής κρίσης. Στη Λιθουανία έχουμε κάνει κάποιες εκτιμήσεις για το ε, πόσο θα μειωθεί το ΑΕΠ μας λόγω του ρωσικού αποκλεισμού στα γεωργικά μας προϊόντα. Και ένα τελευταίο που θα σας παρακαλούσα να κοιτάξετε είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Βεβαίως η Λιθουανία καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για τις ε, συνοριακές διασυνδέσεις. Έχουμε στον Κλέπεντα ένα σταθμό ε, υγροποιημένου φυσικού αερίου ε, που θα ολοκληρωθεί ο τερματικός αυτός σταθμός στα τέλη του έτους. Και θέλω να πω και στους συναδελφούς ότι στη Λετωνία, το ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν φυσικό αέριο και αγωγό και επίσης σε ό,τι αφορά ε, την διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων grid, έχουμε το polling που είναι σύνδεση Πολωνίας-Λιθουανίας. Αλλά και εκεί ανησυχούμε ε, σε σχέση με κάποια έργα που πρέπει να γίνουν από πολωνικής πλευράς και στην πολωνική επικράτεια. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συζήτηση αυτή. Εδώ πραγματικά πρέπει να γίνονται αυτές οι συζητήσεις και να ακούγονται κάποια σχόλια. Ευχαριστώ. Τώρα, από τις κάτω χώρες, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ε, κυρία Σχόχτ. Κύριε Πρόεδρε, στα αγγλικά επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή σας που διοργανώνει αυτή την διακοινοβουλευτική ανταλλαγή απόψεων για να απαντήσουμε για τις βέλτιστες πρακτικές που μας ρωτήσατε στην Ολλανδία. Πρώτον, οι αρμόδιες κοινοβουλευτικέ επιτροπέ θα πρέπει να εξετάζουν τι ευρωπαϊκέ επίση πολιτικέ ε, που είναι θέματα αρμοδιότητά τους στι επιμέρου, Για τι συστάσει αναχώρα για τον προπολογισμό, δημόσια υγεία, τι συντάξεις και την ε, αγορά Στέγη, αυτά συζητώνται στις αρμόδιε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ περισσότερο, στι κλαδικέ και επιμέρου, και όχι στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Επίση, για το πρόγραμμα σταθερότητα και τι μεταρρυθμίσει γίνεται πάντα μια συζήτηση πριν σταλούν τα προγράμματα στις Βρυξέλλες για να μπορεί το Κοινοβούλιο να τα προσαρμόζει. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση ακολουθεί στον προπολογισμό της συστάσης μετά από επεξεργασία από πλευράς Κοινοβουλίου και το τηρεί αυτό αυστηρά. Τώρα για τα σχέδια της κυβέρνησης για το 2015, την προηγούμενη διετία η κυβέρνηση πήρε πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας που οδήγησαν σε μείωση του ελλείμματος από 4,5% που είχαμε του προπολογισμού το 2011 σε 2,8% φέτος. Για το επόμενο έτος δεν προβλέπονται νέες περικοπές στον προϋπολογισμό παρόλο που πολλές από τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις και περικοπές εξακολουθούν να ισχύουν. Ευτυχώς η οικονομία μας βγαίνει σιγά σιγά από την ύφεση φέτος. Για παράδειγμα το κόστος στην υγεία έχει μειωθεί σημαντικά γιατί έχει αποκεντρωθεί η εκτέλεση σε επίπεδο ε, τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι πιο στοχευμένη η ε, περίθαλψη. Όλα αυτά συνάδουν με τις συστάσεις που είχαμε αποτέλεσμα και συμπέρασμα. Ο δείκτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι θετικός και πάλι για την Ολλανδία και δεν είμαστε σε διαδικασία πλέον υπερβολικού ελλείμματος. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα επανερχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει το λόγο Indigo Galpelts από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Επιτρέψτε μου να πω ένα θερμό καλωσόρισε στους ε, εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία να έχουμε τέτοια συνάντηση, να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα και θέλω να συζητήσουμε τα εξής. Καταρχάς να απευθύνω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια θα ήθελα να σχολιάσω την ε, έκθεση. Πολλοί συνάδελφοι θα σημειώνουν ότι υπάρχουν ζητήματα προς την εφαρμογή, την υλοποίηση των ε, συστάσεων ανακράτος, ανακράτη. Ε, και άλλοι λένε ότι η ίδια η σύσταση σαν όρος συνεπάγεται και συνεργασία μεταξύ των δύο εταίρων. Για να είναι αρκετά φιλόδοξη λοιπόν και θα πρέπει να είναι λοιπόν χρήσιμη ε, για τα κράτη αλλά και αρκετά φιλόδοξη η σύσταση ανακράτος. Ωστόσο θα πρέπει να πω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ποτέ υποχρεωτική μια σύσταση ούτε να τιμωρείται κανείς ή να του επιβάλλεται πρόστιμο επειδή δεν υλοποίησε μια σύσταση. Δεν μπορεί με τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα. Άρα χρειάζεται διαφορετική μεθοδολογία. Και όσον αφορά την έκθεση θα ήθελα να συγχαρώ τον συντάκτη τη Έχει πάρα πολύ καλή δομή. Διατυπώνω ωστόσο αρκετέ τροπολογίε, γιατί βλέπω να λείπουν κάποια σημεία. Συμφωνώ δε με τους συναδέλφου που είπαν ότι πολλά μένουν να γίνουν και ότι δεν είναι αρκετά πιστική αυτή η οικονομική ανάπτυξη. Οι δικέ μου τροπολογίε εστιάζονται στην ε, ε, στεναρότητα, τις δυνατότητες και ένα πολύ σημαντικό τομέα ως προς τις, ε, την ισχύ μας που δεν αξιοποιείται επαρκώς. Η, ισχύ μας είναι η εσωτερική αγορά. Πρόκειται για έναν πυλώνα που θα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω. Έχω καταθέσει και τις προτάσεις μου. Ε, και νομίζω ότι εάν ενισχύσουμε περισσότερο την εσωτερική αγορά μπορούμε να συμβάλλουμε στην οικονομική ανάκαμψη, δυνατότητες που υπάρχουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολλές ε, επιχειρήματα που διαρκώς υπογραμμίζουμε και επαναλαμβάνουμε, τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν να κάνουν με την ε, πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση πάνω απ' όλα. αλλά εδώ έχουμε σαν επιπλέον απώλεια, την ε, απώλεια της κοινωνικής συλλογής, την ανεργία, τα σημαντικά προβλήματα στην οικονομία. Όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν, εάν στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα, ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, δηλαδή ένα αλλακτικό σύστημα που θα μπορούσε να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να τα λύσουμε. Έχω αναφερθεί σε θέματα και φορολογία σε μια από τις τροπολογίες μου, που έθιξαν και άλλοι συνάδελφοι λέγοντα ότι είναι εθνική αρμοδιότητα. Σε αυτό συμφωνώ φυσικά, αλλά θα ήθελα ταυτόχρονα να υπογραμμίσω και κάτι άλλο που έχω συμπεριλάβει σε έκθεση για την ε, φορολογία, ότι η φόρο αποφυγή ή η αλλαγή των επιπέδων φορολόγησης πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χρειάζεται να έχουμε πιο πολλές ε, πληροφορίες και γνώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μπαγέ από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίζω και εγώ τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και το συντάκτη της εκθέσεως ε, στην οποία μπορούμε να συμφωνούμε σε πολλά σημεία ασφαλώς αν και σε ορισμένα αρκετά τα σημεία πάλι δεν συμφωνούμε. Θα ήθελα να συνεχίσω στα όσα είπε η ε, συντονίστριά μας ε, Φερέιρα. Ε, μία προϋπόθεση, ένα δεδομένο το οποίο υπογραμμίζεται και το οποίο, στο οποίο εμείς δεν συμφωνούμε που λέτε ότι οι ιδιωτικέ επενδύσεις είναι καλύτερες από τις δημόσιες. Εγώ έχω μια σειρά παραδείγματα να σας αποδείξω ότι έχετε άδικο σε αυτό στις βρετανικές συνδρομικές επιχείρησεις τη σημειώνονται όλο και περισσότερα ατυχήματα. Οι επενδύσεις ιδιωτικέ οι οποίες... Ε, ε, στις τράπεζες σε παραδείγματι έχουν οδηγήσει πολλές φορές σε τεράστια προβλήματα ε, φόρτις και πολλά άλλα που έχουμε από το Βέλγιο. Ε, άρα πρέπει να βρούμε μία ισορροπημένη αναλογία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, παραδείγματι για, τους, ε, για τις βιομηχανικές ζώνες, για τους αυτοκινητοδρόμους, ε, και, σε πολυ... και το... τα πολυλειτουργικά μέσα ασφαλώς είναι πολύ πιο αποδοτικές οι κρατικές επενδύσεις από τις θετικές. Θα υπογραμμίσω επίσης ότι η φλαμανδική κοινότητα αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τον περιφερειακό της Αμβέρσης ακριβώς για να διαφυλάξει την κινητικότητα και την αποτελεσματικότητα στις εργασίες των πολιτών. Αυτό λοιπόν πρέπει να το υπογραμμίσουμε γιατί είναι μια πραγματική επένδυση, δεν είναι λεφτά πεταμένα από το παράθυρο και πρόκειται να καταθέσουμε μια ε, τροπολογία την οποία ελπίζω ότι θα μελετήσετε με μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Τσάραν Λίντς από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, πρόεδρος της Επιτροπής των ε, Δημοσιονομικών. και με συγχωρείτε πρόεδρε που δεν μπορούσα να αφήσω το κουμπί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα βγαίνει σας λόγια. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε σήμερα για να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι η πρώτη φορά όπως ξέρετε που η Ιρλανδία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο χάρη στην επιτυχία ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που ε, σημαίνει ότι η Ιρλανδία έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις και επανήλθε στις αγορές κεφαλαίων το Δεκέμβριο του 2013. Τα τελευταία δεδομένα που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα είναι πολύ ενθαρρυντικά για την Ιρλανδία. Είχε αναθεωρηθεί η πρόβλεψη προς τα άνω για το ΑΕΠ κατά 4,5%. Έχουμε στόχο να ξεπεράσουμε το έλλειμμα του 3% επί του ΑΕΠ έως το 2015. Όταν επιτευχθεί αυτό θα έχουμε επιτύχει έναν στο στόχο συσκελισμένου προπολογισμού όπως αρχικά είχαμε δηλώσει. Όπως καταγράφεται στην έκθεση, ε, το Εθνικό Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει ενεργά στην ε, ε, διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η δική σας Επιτροπή έχει ε, η δική μας Επιτροπή μάλλον των Οικονομικών έχει συνεργαστεί και με το αρμόδιο Υπουργείο πριν από την επεξεργασία και υποβολή των συστάσεων. Ε, αρκετές κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν συζητήσει τα θέματα αυτά με αρμόδιους υπουργούς όπως αυτών της Εθνικής Οικονομίας ενώπιον της Επιτροπής των Οικονομικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην αντίστοιχη Επιτροπή και Έχουμε συζητήσει επίσης τα θέματα όλα αυτά πριν να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του προπολογισμού με τους εμπλεκόμενους φορείς προσπαθώντας να τους υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αναχώρα πριν κατατίθενται οι προτάσεις ε, για τον προπολογισμό. Ε, έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε, να εξετάσουμε τις συστάσεις αναχώρα και να να βεβαιωνόμαστε ότι τηρούνται όπως προβλέπεται ανάλογα με την εφαρμογή του στον κάθε τομέα. Πολλές είναι οι επιτροπέ, οι οποίες συνεχίζουν την παρακολούθηση των προετοιμασ... της προπαρασκευής αυτής της διαδικασίας σε επίπεδο Ιρλανδίας ε, σε συνεργασία και με τους αρμόδιου υπουργούς. Οι συστάσει ανά ε, κράτος είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να προσμετρηθεί το μέγεθος και η απόδοση της οικονομίας και να δούμε εάν τηρούνται τα ορόσημα ω προς τη διακυβέρνηση. Ωστόσο θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το χρονοδιάγραμμα ανάμεσα στη δημοσίευση των συστάσεων αναχώρα και, της, ε, και, την, και της υιοθέτηση από το Συμβούλιο ε, δεν επιτρέπει την εξέταση από την Επιτροπή των Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί περισσότερο χρόνος χρόνο στα Εθνικά Κοινοβούλια για να μελετήσουν τις συστάσεις αναχώρα. Προηγούμενε ε, μελέτες και εξετάσεις αυτών των συστάσεων είχαν δώσει περισσότερο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των συστάσεων ανά κράτος. Αυτό είναι απαραίτητο και νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί μια καλύτερη ευκαιρία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και για τα Εθνικά Κοινοβούλια να συναντιούνται μαζί για να συζητούν τη, στην κατάλληλη χρονική στιγμή βεβαίω τι συστάσει ανακράτο. Επίση, για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι εν γέννη οι αναχώρα έχουν, ε, είναι ιδιαίτερα εύστοχες ως προς την οικονομία της ε, Ιρλανδίας. Η τάση για μείωση του ε, ελλείμματος της χώρας κάτω από το 3% είναι πάρα πολύ σημαντική. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει βεβαίως να συνοδεύεται και θέλω ιδιαίτερο να το υπογραμμίσω αυτό γιατί είναι κάτι που αφορά και την Ιρλανδική Προεδρία. Θα πρέπει να συνοδεύεται και με παραγωγικές, ε, από παραγωγικές επενδύσεις και ιδιαίτερως θέλω να διαρωτηθούμε όλοι μαζί τι σκοπό εξυπηρετεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με την ε, λογοδοσία βεβαίως, με τη δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας και νομιμοποίηση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε σε επενδύσεις, κεφαλαϊκές επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα σχέδια τα οποία θα βοηθήσουν όλες ε, τις χώρες να προχωρήσουν αλλά θα πρέπει αυτό να προσφέρει ένα κοινωνικό μέρισμα γιατί πρέπει να έχουμε ένα ε, μια ειδική σύσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο για την κάθε χώρα όταν βγαίνουμε από την περίοδο της κρίσης σιγά σιγά, πρέπει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα να μην είναι μόνο μια προσπάθεια για ισοσκελισμό των εθνικών προϋπολογισμών, αλλά και μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε τη διαδικασία αυτή της ενοποίησης που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 40. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες στο μοντέλο του εξαμήνου, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ εστιασμένες στις χώρες σε κάθε περίπτωση προσπάθειες, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ε, αναπτύξουμε αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το σχέδιο σε πιο ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ πολύ και τον διακόπτη ομιλητή. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μία σύσταση για την Ευρωζώνη, όχι για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Καμπρίτα που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού και Οικονομία του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ. Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή την ευκαιρία συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων και των εκπροσώπων της ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορέσουμε να σκεφτούμε από κοινού, να προβληματιστούμε από κοινού για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Διότι στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή κρίση αυτό που ε, έλειπε ήταν ο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και η δημοκρατική συμμετοχή που θα νομιμοποιούσε τι αποφάσει που ελήφθησαν για την καταπολέμηση τη κρίση. Γι' αυτό το λόγο ε, και δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του αποτελεί ένα βήμα στη θετική κατεύθυνση για καλύτερο συντονισμό και διασύνδεση των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη συμμετοχή των όσων αντιπροσωπεύουν, είναι δηλαδή ερετοί, των ευρωπαϊκών ε, λαών. Γι' αυτό και θα πρέπει εδώ να συζητήσουμε ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτό το συντονισμό, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η Ευρώπη βρίσκεται στην όχθη, στο χείλος του αποπληθωρισμού με μηδενική ανάπτυξη σχεδόν και με δημοσιονομική εξυγένση που σε πολλές χώρες δεν είναι διόλου φίλοι με το, την ανάπτυξη. Στην Πορτογαλία ακριβώς αυτό ζούμε. Μόλις βγήκαμε από τρία χρόνια πολιτικών αναπροσαρμογών ε, και συνοδεία της Τρόικας ε, και ε, είδαμε την αύξηση του δημοσιογράφου στο 40% του ΑΕΠ, τρία χρόνια λοιπόν μεταρρυθμίσεων και στρατηγικές επιχειρήσεις για την πορτογαλική οικονομία χάσαν τις διαστάσεις τους, αποσυντέθηκαν, διαλύθηκαν, φτώχευσαν χάσαν τις δυνατότητες συμβολής στην ανάπτυξη της χώρας και ε, γι' αυτό τον λόγο η Πορτογαλία δεν έχει λάβει συγκεκριμένες συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου γιατί τούτη η Επιτροπή στις αρχές της εντολής αυτή, το, αυτής της θητείας του Κοινοβουλίου εκμεταλλεύτηκε τα συμπεράσματα ε, τη, των όσων έκανε η Τρόικα το τελευταίο χρονικό διάστημα και αποφάσισε να προβληματιστεί για το τι, ποια ήταν τα αποτελέσματα του συντονισμού. Σε αυτά τα πλαίσια το να βρεθούν τρόποι συντονισμού λοιπόν που θα επιτρέψουν τη συνδυασμό το δημοσιονομικής ε, πολιτικής με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτά τα απαραίτητα στοιχεία για τον ε, δημοσιονομικό συντονισμό, δηλαδή η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, η αποφυγή της διαφυγής κεφαλαίων σε φορολογικούς επανδύσεις ακόμα και εντός της Ευρωζώνης ή με την κατάσταση επιχειρήσεων ε, και να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στην τραπεζική Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε τους μηχανισμούς εγγύησης των καταθέσεων. Μέσα σε αυτή τη μεταρρύθμιση λοιπόν που είναι δυναμική και που θα πρέπει να διέπει την αυξανόμενη συντονισμό των οικονομικών πολιτικών για να έχει νόημα τόσο για το μέλλον της Ευρώπης όσο και για την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και γι' αυτό το, ευρωπαϊκό, το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο θα είναι πάντα ανοιχτό στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευρωβουλευτές τώρα, ο Μπέντ Λούκε από το ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Ich würde jetzt gerne an dieser... ναι, εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της Γερμανικής Βουλής ε, ή ακόμα και κάποιο διοικητικό υπάλληλο θα επιθυμούσα, δυστυχώς απουσιάζουν άπαντες. Λάμπει δια της απουσίας του η Γερμανική Βουλή. Αυτό το βρίσκω πάρα πολύ λυπηρό, είναι και προσβολή πιστεύω ε, προς την Επιτροπή μας, γιατί συμφωνούμε όλοι ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι σημαντικό μέτρο για τις οικονομικές πολιτικές, για να συνοδεύονται από συστάσεις που τα κράτη-μέλη, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Και εδώ θα έπρεπε να ακούσουν τα μέλη της Μπούντεστα και να τοποθετηθούν. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό και ενοχλητικό γιατί η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται ούτε για τα μάτια δεν ε, υποδίεται ε, ότι ε, λαμβάνει τουλάχιστον υπόψη της τις συστάσεις. Θυμίζω ότι ε, γίνεται λόγος για απλούστευση και μεταρρύθμιση των φορολογικών συστημάτων με διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Στη Γερμανία δεν το βλέπουμε αυτό πουθενά. Δεν υπάρχει νομοθετική τέτοια πρωτοβουλία ούτε εγχείρημα. Πρέπει να αλλάξει το επίδομα ε, μητρότητας γιατί τώρα ε, επιβαρύνει ιδιαίτερα τα ασφαλιστικά ταμεία. Από ό,τι φαίνεται ούτε αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη, ούτε καν γνώση του η κυβέρνηση. Επίσης ε, γίνεται λόγος για αύξηση και όχι μείωση του όριου συνταξιοδότησης. Ε, και, η γερμανική κυβέρνηση δεν αυξάνει το αλλά προτείνει 63 έτη. Επίσης, σύνταξη θα πρέπει να ενισχυθεί ε, και πάλι τίποτα δεν κάνει εκεί. Και είναι πολύ δύσκολο να ενισχυθεί η διαδικασία κεφαλαιοποίησης εάν ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, οδηγεί σε μια πολιτική ε, με τεράστια συμπίεση των επιτοκίων οπότε δεν συμφέρει να ε, αποταμιεύει κανείς χρήματα. Όλη αυτή την κριτική από ό,τι φαίνεται ε, δεν τη λαμβάνει υπόψη καθόλου ε, η Γερμανική Βουλή η οποία σύμπασα απουσιάζει εδώ. Και ένα τελευταίο, οι συστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται και επί της ουσίας κατά πόσο είναι συνεκτικές και συνεπείς με την ουσία. Γιατί από τη μια ζητούν από τη Γερμανία να μειωθούν οι φόροι και από την άλλη, για παράδειγμα, ζητούν ε, τα επιδόμετα ε, ε, μητρότητας να χρηματοδοτούνται από τους κρατικούς πόρους, άρα αύξηση φόρων. Τέτοιες στάσεις δεν είναι σκόπιμες ούτε εύστοχες και θα πρέπει να συνάδουν αυτά που προτείνουμε με τα όσα καλούνται να υλοποιήσουν οι χώρες. Ευχαριστώ. Η Ντανούτα Χούβνερ, παρακαλώ. Uh, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια στο πλαίσιο των τροπολογιών που εγώ και η ομάδα μου καταθέσαμε. Ανέφερθηκαν ήδη από την Ιβάνα Μάλετιτς. Ίσως θα θυμάστε ότι όταν διαπραγματευόμασταν ως κοινοβούλιο για το, την πολιτική συνοχής και το πλαίσιο της για το 2014 μέχρι το 2020, θελήσαμε να εισάγουμε μέτρα τα οποία συνδέουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο μέσων με την στιβαρή οικονομική διακυβέρνηση και συγκεκριμένα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαμε εδώ για το θέμα της πιο βαθιάς και πιο αποτελεσματικής χρήσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου, Διευθυντικού Ταμείου για να στηριχθούν οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και οι επενδύσεις που χρειάζονται σήμερα για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να βγούμε από την κρίση και Το θέμα αυτό επανήλθε εδώ και καιρό. Επανέρχεται μάλλον εδώ και καιρό. Και αυτή η σχέση ανάμεσα στα ταμεία και το ευρωπαϊκό εξάμεινο τα έχουμε στη διάρκεια της πολιτικής συνοχής ενώ προσπαθούμε να φτιάξουμε εταιρικέ σχέσεις με, και συνεργασίες με τα λειτουργικά προγράμματα για τις συγκεκριμένες συστάσεις για τα κράτη-μέλη. Ανά χώρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή νομίζω να εξασφαλίσουμε πως υπάρχει αυτή η σύνδεση και θα γίνει η πραγματικότητα ώστε να έχουμε στήριξη όχι μόνο για τις δημόσιες επενδύσεις, αλλά ξέρουμε ότι τα, η δραστηριοτική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση διευκολύνει τη χρήση και προσκαλεί, προσελκύει τις ιδιωτικές επενδύσεις στο σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να προσθεθεί φέτος στις συστάσεις αναχώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Τώρα, ο Ζόρζο Κιλζινέ από το Βελγικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση τη σημερινή. Πιστεύω πως ο διάλογος ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο είναι απαραίτητος αλλά θα πρέπει να εντατικοποιηθεί περισσότερο. Τα τρία λεπτά αγόρευση, χρονομιλίες που έχουμε δεν αρκούν για να λυθεί το θέμα της νομιμότητας από τη μια πλευρά ανάμεσα στις συστάσεις της Κομισιόν και από την άλλη πλευρά την αυτονομία των κρατών και την πολιτικές επιλογές. Είμαι Ευρωπαίος βεβαίως 100% αλλά θα ήθελα ο διάλογος να επιτρέψει ε, προσαρμογές και από τις δύο πλευρές, από τα Εθνικά Κοινοβούλια να μπορούν να έχουν ακόμη περισσότερο λόγο σε σχέση με τις συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη. Αυτό για τη διαδικασία. Ήδη υπάρχει βέβαια πρόοδος γιατί είμαστε εδώ και συνομιλούμε. Επί της ουσίας η βασική επίκριση που θα είχαμε να διατυπώσουμε είναι το θέμα του ρυθμού της επιστροφής στην δημοσιονομική ισορροπία και πειθαρχία που συνδέεται άμεσα με την λειτουργία της οικονομίας μας. Πώς θα εξηγιανθεί η εθνική οικονομία χωρίς να στραγγαλιστεί η οικονομική δραστηριότητα. Πώς θα κάνουμε για να επενδύσουμε στα κράτη, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για το μέλλον, πώς να διατηρηθούν όμως ταυτόχρονα οι δαπάνες για τα κοινωνικά θέματα που εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και την εσωτερική κατανάλωση που κάνει την οικονομία, τις οικονομίες μας να δεκινούνται. Πώς θα δούμε λοιπόν τις συνέπειες. Οι συνέπειες για τη κράτη και για τις ε, βελγικές περιφέρειες είναι πολύ συχνά η μείωση των επενδύσεων ή ε, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που πονάνε και που κάνουν τους πολίτες να χάνουν την εμπιστοσύνη τους ε, στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνω για επιτριών ε, θεμάτων που πιστεύω πως δεν ε, αντιπροσωπεύονται επαρκώς. Πρώτος άξονας είναι ο άξονας της ενέργειας, της, ε, ε, ε της ενεργειακής επάρκειας, της αναζήτησης οικονομιών. Είναι πολύ θεμελιώδες θέμα ε, και στρατηγικό. Το βλέπουμε σε σχέση με τη Ρωσία, το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά και από οικονομικής άποψης δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε σήμερα το θέμα της ενέργειας από το θέμα το δημοσιονομικό. Ε, θα έπρεπε να είναι λοιπόν πολύ πιο παρόν το θέμα αυτό στις συστάσεις. Δεύτερο στοιχείο είναι το κοινωνικό, όπου πιστεύω ότι αντί για μείωση με κάθε κόστος του κόστους της εργασίας ε, θα πρέπει να αναζητήσουμε περισσότερη κοινωνική σύγκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μπορέσουμε να ε, διερωτηθούμε όσον αφορά τις συνέπειες της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Είδαμε τη λέξη προστατευτισμός, υπάρχουν κάποιες μορφές προστατευτισμού, αλλά σίγουρα η πρόοδος δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των οικονομιών άλλων, γιατί διαφορετικά καταλήγουμε σε ασυνεννοησία ανάμεσα στους εργαζόμενους και πρέπει να αναζητηθούν τρόποι με την της οικονομίας που θα δαπανά λιγότερο μάλλον που θα εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, αλλά θα ευνοεί ε, τις νέες επιχειρήσεις. Έπειτα πιστεύω πως η Κομισιόν είναι πιο λιγότερο σκληρή απέναντι στα χρηματοπιστωτικά συστήματα από ό,τι απέναντι στα κράτη. Πρέπει ναι, να μεταρρυθμιστεί το τραπεζικό σύστημα αλλά και να προσανατολιστεί στην πραγματική οικονομία, δάνεια στις επιχειρήσεις μας και όχι στους κερδοσκόπους. Θα πρέπει δηλαδή να βελτιωθούν τα βασικά στοιχεία ε, για την καταπολέμηση της φοροαπάτης και συμβολή στην επιστροφή στην δημοσιονομική ισορροπία με το φόρο, για παράδειγμα, ε, των ε, επιτών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δηλαδή, ε, κοινωνικά θέματα, ενέργεια και οικονομία. Θα πρέπει περισσότερο να, είναι στη τελική, να τονίζονται στη τελική έκθεση. Ευχαριστώ. Το, το λόγο έχει ο Καμπριέλε Ταμάντο που είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού του Αυστριακού Κοινοβουλίου. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα μιλήσω και εγώ γερμανικά. Ευχαριστώ για την ε, πρωτοβουλία να μας καλέσετε εδώ για ανταλλαγή απόψεων από αυτού του θέματος. Στην Αυστριακή Βουλή μας απασχολούν οι συστάσεις αναχώρα και τις εξετάζουμε ήδη. Ε, υπάρχει και ένα ε, ειδικό συμβούλιο από τον Νοέμβριο του 2013 που ασχολείται με αυτά τα δημοσιονομικά θέματα και επαγρυπνεί κατά πόσο τηρούμε ε, τους κανόνες για τα δημοσιονομικά. Αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκδίδει μια ετήσια έκθεση και την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε για αυτήν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Γίνεται δημόσια δηλαδή η συζήτηση αυτή και ε, αν θέλουμε να παίρνουμε σοβαρά τον εαυτό μας ως εθνικοί βουλευτές, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ορισμένες συστάσεις, για να μην πω πολλές, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες είναι γνωστές ως αδυναμίες, ας πούμε, στις μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος ε, στην Αυστρία ή υπερβολική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας. Το 2013, το φθινόπωρο, είχαμε όπως γνωρίζετε βουλευτικές εκλογές και τώρα ε, στο κυβερνητικό πρόγραμμα ελήφθησαν μέτρα όπου ε, ε, εξομοιώνεται ε, η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ε, με την ε, νομοθετική, γιατί ξέρετε είναι διαφορετική σε ό,τι αφορά τους άνδρες και τις γυναίκες. Οι άνδρες στα 65, οι γυναίκες στα 60. Και πρέπει να εναρμονίσουμε τις δύο ηλικίε και νωρίτερα από ό,τι σκοπεύαμε. Πολιτικά αυτό το θέμα είναι πολύ επίμαχο όμως και η συζήτηση γενικότερα που αφορά αυτά τα ζητήματα, αλλά βέβαια θα πρέπει αντίστοιχα και η αγορά εργασίας ε, να έχει τη δυνατότητα απορρόφησης όλων αυτών των ανθρώπων για να μπορεί να απασχολεί και να εργοδοτεί ηλικιωμένες γυναίκες. Επίσης, επενδύουμε στην ενεργή αγορά εργασίας. Στον προπολογισμό του 2014 έχουμε προβλέψει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας αυτό. Παρ' αυτά, ε, παρά το γεγονός ότι έχουμε το χαμηλότερο δίκτυο ενεργείας στην Ευρώπη, αυξάνεται και σε εμά η ανεργία ονομαστικά και φτάνει στις 400.000, 400.000 ανέργους προσπαθούμε να εξηγάνουμε τον προπολογισμό μας, να τον ισοσκελίσουμε. Έχει συσταθεί από την κυβέρνηση και ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων για να ανταποκριθεί στη σύσταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ελαφρυνθεί από την υπερβολική επιβάρυνση η εργασία. Κάποιοι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και ορισμένοι ευρωβουλευτές είπαν ότι οι συστάσεις έχουν και πολιτική διάσταση και ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να λαμβάνουν ε, κυρίαρχα τις πολιτικές τους αποφάσεις. Προφανές είναι αυτό. Και για μας ε, είναι μια συζήτηση αυτή που γίνεται και επανέρχεται. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να βελτιώσουν και τη λειτουργία τους και τη συνεργασία τους για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των βουλευτών, συνεδριάσεις κοινοβουλευτικές για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά και αλληλογραφία. Δηλαδή έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συστάσεις προς ε, τις κυβερνήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω και αυτή η επικοινωνία χωράει βελτίωση και ο συντονισμός. Πάντως στην Αυστρία πέρα από κομματικά όρια έχουμε συμφωνήσει ε, για την ενεργή συνεργασία μας σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Μαριάς. Ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια στη συνεδρίασή μας και βέβαια να επισημάνω ότι δεν υπάρχουν ε, Έλληνες βουλευτές, δεν υπάρχουν μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και το με το Προεδρείο. Όπως επίσης δεν υπάρχουν, όπως είπε και ο συνάδελφος κύριος Λούκε, και βουλευτές από τη Γερμανία. Εγώ δίνω εξηγήσει που έχουν άμεση σχέση και με τα δύο. Διότι μεν βουλευτές από τη Γερμανία αισθάνονται, όπως είπε και ο κύριος Λούκε, ότι μπορούν με τις αποφάσεις που παίρνουν στο κοινοβούλιο τους, αλλά κυρίως με την πολιτική που ασκεί η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε, να επιβάλλουν την πολιτική τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για δε την Ελλάδα είναι δεδομένο ότι οι αποφάσεις που παίρνονται στο ελληνικό κοινοβούλιο υπαγορεύονται και επιβάλλονται από την Τρόικα. Επιβάλλονται από τους δανειστές και επομένως η όποια συμμετοχή τους εδώ αντιλαμβάνομαι ότι θα επιβεβαίωνε για άλλη μια φορά αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές στην Ελλάδα και το έχω πει και εγώ σαν βουλευτής. Ότι σήμερα στην Ελλάδα η οικονομική πολιτική που ασκείται επιβάλλεται από την ίδια την Τρόικα και ας έρθουμε στο ίδιο το σύστημα των συστάσεων. Δεν υπάρχουν συστάσεις εξειδικευμένες για την Ελλάδα, για το εξάμεινο, διότι αναφέρεται ότι θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις του μνημονίου. Δηλαδή οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί από τους δανειστές και οι οποίες έχουν οδηγήσει, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε πλήρη οικονομική καταστροφή της χώρας μας. Μάλιστα, το μνημόνιο σύμφωνα με, με απάντηση που έδωσε η Επιτροπή σε συναδέλφους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν σχετική ερώτηση δεν δεσμεύεται από τη Σύμβαση και το Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή είπε η Επιτροπή ότι μπορεί να εφαρμοστεί μνημόνιο στην Ελλάδα παρότι αυτό παραβιάζει τις ίδιες τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει και το Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχουν φτάσει οι χώρες που βρίσκονται στο μνημόνιο. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο επίπεδα. Χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία που επί του πρακτέου είναι εκτός έλεγχο και χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή παλαιότερα η Ιρλανδία ή επίσης η Πορτογαλία οι οποίες έχουν υποστεί τις καταστροφικές συνέπειες των μνημονίων. Διότι με την πολιτική της λιτότητας δεν οδηγούμαστε πουθενά. Υπάρχει τεράστια ανεργία. Στην Ελλάδα έχουν έρθει 214 δισεκατομμύρια ευρώ ως δάνεια και όμως η Ελλάδα έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Το χρέος πλέον έχει ξεφύγει και είναι πάνω από το 175% του ΑΕΠ. Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν υποστεί ζημιά 80 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω του μνημονίου. Η χώρα μας έχει φτωχοποιηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε σε σχέση με τη λειτουργία της Τρόικας και των μνημονίων και επομένως το περίφημο εξάμεινο το ευρωπαϊκό όπου συντονίζονται και συζητούνται οι πολιτικές στην πράξη δεν ισχύει. Στην πράξη γίνεται αυτό που θέλει η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε. Αυτά θεσμικά πρέπει να αλλάξουν και επί της ουσίας η πολιτική της λιτότητας πρέπει να σταματήσει. Now, next speaker, Cora ε, Van Neuer um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της ίδιας της έκθεσης γιατί ο Φίλιπ Τεμπάκε συνάδελφος έκανε εξαιρετική δουλειά από αυτού. Θέλω μόνο να απευθυνθώ στα μέλη των, των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι σήμερα εδώ. Θέλω να σας συγχαρώ που ήρθατε. Είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μοιραζόμαστε μεταξύ μας τις καλύτερες πρακτικές. Νομίζω πως τα θέματα που συζητάμε είναι εξαιρετικά σημαντικά και τόσο μάλιστα σημαντικά που θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα συζητάμε ας πούμε ε, το, ε, τις συστάσεις αναχώρα, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να βλέπουμε πώς εφαρμόζονται στα, στις διάφορες χώρες. Ε, όπως ήδη ανέφεραν οι συνάδελφοι, ε, δεν, δεν έχει εδώ ε, Γερμανούς ούτε Έλληνες εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά πολύ σοβαρό είναι το γεγονός ότι λείπουν και άλλοι συνάδελφοι από άλλε χώρε. ελπίζω, και μάλλον πέρυσι όταν ήμουν εδώ και μίλησα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ εξ ονόματο του Εθνικού μου Κοινοβουλίου, ήταν τα ίδιο, το ίδιο. Πολλές χώρε λείπαν. Ε, κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι κάποιες χώρες που λείπουν δεν βρίσκουν τα θέματα μα σημαντικά. Ε, δεν έχουν κάποια καλύτερη πρακτική να μοιραστούν μαζί μας, αμφιβάλλω. Ελπίζω να μην είναι αυτό. Και κάτι πρέπει να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Πριν από μια ώρα λάβαμε ένα φυλάδιο από την Διεύθυνση Επαφών με την Εθνικά Κοινοβούλια, τον δικό μας εταίρο για την συνεργασία. Πολλά πρέπει να γίνουν εδώ λοιπόν, ίσως του χρόνου να είναι όλες οι χώρες εδώ και θα ήθελα να ζητήσω από τους εθνικούς βουλευτές ε, στις πολιτικές τους ομάδες ίσως να δουν ε, και με τους συναδέλφους από άλλες χώρες γιατί δεν έρχονται και τι μπορούμε να κάνουμε για να επιτύχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή του χρόνου. Ευχαριστώ. Now, ε, the Στραν Τζουρτοβίτς από το κρατικό κοινοβούλιο, πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού και Οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή τη σχέδια έκθεση, Πιστεύω πως πραγματικά έχει περιλάβει τις περισσότερες πτυχές που ενδιαφέρουν τα Εθνικά Κοινοβούλια η πλήρη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, είναι κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και καιρό και για άλλη μια φορά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως αυτό θα πρέπει να γίνει πληρέστερα μέσω επαφών και αναλύσεων ε, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάτι το οποίο βλέπουμε στην έκθεση αυτή που έχει σχέση με το γεγονός ότι μόνο 10% των συστάσεων συγκεκριμένων μάλλον συστάσεων αναχώρα εφαρμόστηκαν πλήρως. 45% των συστάσεων εφαρμόστηκαν μόνο σε περιορισμένο ε, βαθμό. Αυτό είναι πολύ βασικό για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται σε οικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο. Ακόμα και αν έχουμε δηλαδή πολύ καλές αποφάσεις ή συστάσεις, εάν δεν εφαρμόζονται δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχουμε αποτελέσματα εάν δεν εφαρμόζονται. Οπότε, πώς καταλαβαίνετε, χωρίς εφαρμογή τίποτα από όλα αυτά δεν έχει σημασία. Τώρα, όσον αφορά την Κροατία. Έχουμε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η Κροατία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ε, επικρατούσε ύφεση και πρέπει να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε ορισμένους τομείς που εδώ και κάποια χρόνια ε, βρίσκονται σε ύφεση όπως ο κατασκευαστικός τομέας. Οι συστάσεις δεν αρκούν λοιπόν, χρειάζεται περισσότερη συνεργασία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε. Ευχαριστώ Μακάρτα. Να καλωσορίσω και πάλι ε, τους εκπροσώπους των κρατών μελών και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή της έκθεσης. Από προσωπική μου άποψη ε, θέλω να ευχαριστήσω τον, ε, την Μαρίζα Ματίας που διατέλεσε σκιώδης εξ ονόματος της GUNGL και που επέβαλε κάποιες τροπολογίες που νομίζω πως εάν γίνουν αποδεκτές θα καταστήσουν πολύ πιο ισχυρό αυτό το έγγραφο προβληματισμού. Ένας από τους συναδέλφους νωρίτερα μίλησε για την ισορροπία ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά όταν ε, ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Εγώ πιστεύω πως είναι πιο ουσιώδης η δυσκολία, ότι δηλαδή υπάρχει απόλυτο δημοκρατικό έλλειμμα στο επίκεντρο αυτής της δικασίας. Έχουμε διάφορα κρατημέλη που εκπροσωπούνται εδώ από τους εθνικούς τους εκπροσώπους, αλλά διερωτώ με πόσοι από τους ε, ε, ψηφοφόρους τους, ε, οι πλούσιοι τους γνωρίζουν καν ότι γίνεται τέτοια συνεδρίαση. Ακόμα και όλοι οι βουλευτές, οι εθνικοί βουλευτές δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοιες επαφές. Η πραγματικότητα των όσων ακούστηκαν ε, είναι όσον αφορά δηλαδή την οικονομική ανάκαμψη είναι παραπλανητική ε, ε, για τις χώρες ε, όπου υπήρξε κρίση όπως στην Ιρλανδία αυτοί που ήταν στη χειρότερη θέση είναι ακόμα σε, σε πολύ χειρότερη θέση σήμερα ενώ υποτίθεται η χώρα βγήκε από την κρίση οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν πως έχουν φτωχύνει ακόμα περισσότερο τώρα και πολλές περιφέρειες εντός των κρατών μελών όπως το δική μου χώρα έχουν υποφέρει δυσανάλογα ως αποτέλεσμα των μέτρων που εισήχθησαν. Και αυτό ε, πάλι ε, παραπέμπει στο έλλειμμα το οποίο ανέφερα και στην αρχή. Θα ήθελα να παροτρύνω όλους να σκεφτούν ε, σε σχέση με τις ειδικές συστάσεις αναχώρας. Κάνουμε κάτι πιο ριζοσπαστικό. Ας εισάγουμε μια διάταξη ότι καμία σύσταση ειδική αναχώρα δεν θα μπορεί να υιοθετηθεί από μια κυβέρνηση αν έρχεται σε αντίθεση με εκλογικές υποσχέσεις που ε, κανέναν πριν από εκλογική περίοδο. Νομίζω πως ε, θα πηγαίναμε πολύ καλύτερα έτσι, γιατί το θέμα ε, δεν είναι αν είναι υπόλογοι στο Ευρωπαϊκό ή στο Εθνικό Κοινοβούλιο οι βουλευτές. Οι περισσότεροι, όλοι εκλέγονται από τους λαούς. Πρέπει να είναι υπόλογοι στους λαούς τους, στους πολίτες των κρατών μελών. Εγώ λοιπόν αυτό που ήθελα να ζητήσω να κάνουμε όλοι μαζί είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα, μέτρη, τα μέτρα μάλλον θα κινητοποιήσουν τις τοπικές οικονομίες και θα ε, δώσουν αυτές τις επενδύσεις που θα επιτρέψουν σε όσους ε, επηρεάστηκαν πολύ αρνητικά ως αποτέλεσμα των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων που συνεχίζουν να επιβάλλονται ως αποτέλεσμα αυτής της ομαδικής ε, προσπάθειας ε, να δούμε ότι αν λειτουργεί αυτή η οικονομική ε, μεταρρύθμιση. Δεν λειτουργεί για τους περισσότερους και οι πιο αδύναμοι χρειάζονται στήριξη. Και τώρα ο κύριος Ζαριανόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από όσα είπε χθε ο κύριος Δράγκη, αλλά και τις σημερινές κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ένα συμπέρασμα βγαίνει η σημερινή πολιτική από την οποία δυστυχούν οι λαοί της Ευρώπης θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί. Όσοι έλεγαν ότι ο κύριος Ντράκη κόντρα δίθεν στην κυρία Μέρκελ εισηγούνταν χαλάρωση, διαψεύστηκαν ή κοροϊδεύουν. Συνεχίζεται η μόνιμη εποπτεία, τα μνημόνια διαρκείας, η επιμονή στο σύμφωνο σταθερότητας, οι αναδιαρθρώσεις με ένα κέντρο, την τιμή, την μείωση της τιμής εργατικής δύναμης. Χαλάρωση υπάρχει, αλλά μόνο για τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε λίγες μέρες μόνο τους δόθηκαν 82 δισεκατομμύρια ευρώ και συνεχίζεται ο πακτολός δωρεάν χρήματος. Και από πού θα πληρωθούν αυτά? Όπως λέει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, από τη μετατόπιση των φόρων από την εργασία στην κατανάλωση, δηλαδή περισσότεροι φόροι στους λαούς περισσότερη κατεδάφιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης, κατάρριξη των συλλογικών συμβάσεων και μισθή πείνας. Αυτά λέει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Περικοπή αντιπαραγωγικών κρατικών δαπανών, είπε ο κύριος Δράκη, δηλαδή λιγότερα στην υγεία, στην παιδεία, στο δημόσιο. Τελικά, κάθε μείγμα της ίδιας αυτής πολιτικής, είτε δημοσιονομική πειθαρχία ή χαλάρωση, είτε περιοριστικό είτε επεκτατικό, βάζουν στο στόχο τους τους λαούς. Γι' αυτό άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλούν τις κυβερνήσεις να κάμψουν τις λαϊκές αντιδράσεις στις χώρες με ένταση της κρατικής καταστολής κατά των αγώνων γιατί ξέρουν αυτή η πολιτική δεν φτιάχνεται, δεν διορθώνεται. Μόνο να ανατρέπεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ παρακαλώ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, μια εισαγωγική παρατήρηση και τέσσερα σημεία έχω. Εισαγωγική παρατήρηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε εδώ. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να είναι ενισχυμένη, ε, διαρθρωμένη και διαρκής και να μην αφορά μόνο το ευρωπαϊκό εξάμεινο, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε στη Ρώμη μία διάσκεψη του άρθρου 13 και έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε στα οικονομικά και δημοσιονομικά και δεν βασίζονται στο κοινοτικό δίκαιο, χρειάζεται συντονισμένη κοινοβουλευτική δράση οπωσδήποτε. Και στόχος να μην είναι ποιος παίρνει κάτι από κάποιον άλλον, αλλά πώς αντιλαμβανόμαστε την κοινή μας ευθύνη και υπευθυνότητα για ένα κοινό ευρωπαϊκό στόχο. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση τώρα. Ποια είναι η αφετηρία, γιατί μας διαφεύγει λίγο αυτό, είναι παράλληλο. Έχουμε ένα κοινό νόμισμα, έτσι. Και είμαστε η μόνη κοινότητα που διαθέτει κοινό νόμισμα αλλά ούτε κοινή οικονομική πολιτική, ούτε κοινή δημοσιονομική πολιτική, ούτε κοινή φορολογική πολιτική. Και αν θέλουμε να εξαγάγουμε τα διδάγματα από την κρίση και όχι απλώς να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση, θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα κοινό συντονισμό της οικονομίας του προϋπολογισμού και της φορολογίας σε κοινοτικό επίπεδο. Και έρχομαι λοιπόν στο δεύτερο τώρα σημείο το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Το six-pack, το two-pack, ο μηχανισμός σταθερότητας, η τρόικα κτλ. Είναι μόνο βοηθητικές κατασκευές σε μεγάλο βαθμό διακυβερνητικές με αποδυνάμωση και των εθνικών κοινοβουλίων αλλά και του ευρωπαϊκού συνδέονται. Και η διάρκεια τους επιτρέπεται να είναι μόνο τέτοια μέχρι να αλλάξει η συνθήκη με αναθεώρηση για να ε, βασιστούν όλοι αυτοί οι θεσμοί στο κοινοτικό δίκαιο και να κατοχυρωθούν στη συνθήκη. Όλα αυτά είναι διάμεσες λύσεις που συζητούμε, με Σοβέζικη. Και γι' αυτό σας ζητώ το εξής. Και η Τρόικα θα πρέπει να κατοχυρωθεί και ε, ο μηχανισμός σταθερότητας ο ευρωπαϊκός και έχω και πολύ μεγάλες επιφυλάξεις μέχρι που το απορρίπτω αυτή τη στιγμή να γίνεται μια απόπειρα ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας να εξαιρεθεί, να καταργηθεί αντί να μεταξελιχθεί σε ένα γνήσιο και ουσιαστικό ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο. Μόνο εάν ιδρύσουμε και βασίσουμε στο κοινοτικό δίκαιο ένα ευρωπαϊκό πλέον νομισματικό ταμείο, τότε και μόνο τότε θα έχουμε την πολιτική αξιοπιστία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανα πάσα στιγμή μπορεί να λαμβάνει σταθεροποιητικά μέτρα για ένα νόμισμα, σε περίπτωση που γνωρίζει κάποιες δυσκολίες και προβλήματα. Τρίτο, περιεχόμενο και ουσία. Για το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο. Θυμίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα είναι αρμόδιος και ο κύριος Μοσκοβισή και η κυρία Μαριάν Τέισεν. Οπότε η ανάπτυξη, η απασχόληση, ο υπολογισμό, το νόμισμα, τα κοινωνικά και η εργασία συνδέονται. Και αυτό είναι το πακέτο των κριτηρίων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Για την κοινή λοιπόν δημοσιονομική πολιτική, για να μην γελιόμαστε, και το τέταρτο είναι η εφαρμογή. Πολύ ξεκάθαρα. Οι συστάσεις πρέπει να γίνουν δεσμεύσεις υποχρεωτικές που να συναντεύονται με κυρώσεις. Όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αβίαστα ε, δήλωσαν ότι οι κυρώσεις ε, θα πρέπει να συνδέονται με τις υποχρεώσεις στις οποίες θα έχουν μεταξελιχθεί οι συστάσεις υποχρεωτικά. Διότι η εφαρμογή είναι ανεπαρκής και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις δύο πλευρές με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας Μαυρίδης τελευταίος και μετά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας. Παρακαλώ. Uh, θα ήθελα καταρχάς και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή και όλους τους άλλους που έχουν συμβάλει σε αυτήν την έκθεση. Πρόεδρε, είναι δύσκολο να μιλάμε για οικονομικά θέματα χωρίς να αναφερόμαστε και ιδεολογικά και στο ιδεολογικό περιεχόμενο. Σε αυτό θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ, σε ένα μόνο σημείο δηλαδή, και θα προσπαθήσω να είμαι στο δυνατόν λιγότερο ιδεολόγος. Σε σχέση με τις συστάσεις αναχώρα λοιπόν θα περίμενα να δω πέντε λόγια για το θέμα του ιδιωτικού χρέους, ιδιαίτερα για τα κράτη εκείνα τα οποία έχουν τεράστιο χρέος οφειλόμενο στο τραπεζικό σύστημα. Το επίπεδο του τραπεζικού χρέους, του ιδιωτικού χρέους σε χώρες της Ευρωπαϊκής και περιφέρειες όπως στη Ισπανία, η δική μου η πατρίδα η Κύπρος, έχει τόσο μεγάλη, ε, είναι τόσο δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την ε, συρρήκνωση του ειδικού εισοδήματο που έχουμε τράπεζες ζόμπι. Και χρειάζεται για τους ανθρώπους, να, για τους πολίτες, να δώσουμε μια επιπλέον ευκαιρία, μια άλλη ευκαιρία, μια ειδική λοιπόν σύσταση ευρωπαϊκή, η οποία θα ε, αλλάξει τα πράγματα. Μια λογική εξήγηση για το ότι δεν αντιμετωπίστηκε το ζήτημα, θα μπορούσε για μένα να είναι το ότι ίσως αυτοί οι οποίοι καταγράφουν τις συστάσεις αναχώρα θεωρούν ότι έχει μηδανικό υπόλοιπο το εγχείρημα, ότι δηλαδή όποτε διαγράφεται ένα ευρώ χρέους κάποιος θα πρέπει να το πληρώσει. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με συνήθεις καταστάσεις και συνθήκες. Το να διορθωθεί λοιπόν ένα τέτοιο ζήτημα μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική μέσα στην οικονομία η οποία θα προσθέσει πιστεύω ε, αξία και γι' αυτό υπογραμμίζω την ανάγκη της θεμελί, των θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων της ε, αφαιρεγγιότητας και της ε, πτώχευσης των τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι έχουμε και αντίστοιχη πρόταση από τον Brian Hayes που ίσως θέλει να την επαναλάβει γιατί δεν σημειώθηκε ε, λεπτομερώς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω, θα είμαι σύντομο βεβαίω και καλωσορίζω το διάλογο με όλου του συναδέλφου από όλα τα εθνικά κοινοβούλια και συμφωνώ με του λοιπού συναδέλφου ότι δεν θα πρέπει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο περαιτέρω διάλογος σε όλα τα θέματα. Ιδιαίτερα θέλω να υπογραμμίσω το εξή ότι οι συστάσεις κράτος και η διαδικασία του εξαμήνου που συστήσαμε με βάση την έκθεση Ντεμπάκρη πριν από δύο εβδομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο ε, μπορεί να έχει πραγματικά αποτελέσματα εάν τα κράτη ε, υιοθετήσουν ενστερνιστούν τις τάσει αυτές και τις υλοποιήσουν στην πραγματικότητα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα. Παραδείγματι, γιατί η ανεργία των νέων στη Γερμανία και την Αυστρία είναι κοντά στο 6 και το 7%, όταν είναι 25% στη Βρετανία και την Ιρλανδία. Τι είναι αυτό που κάνουν οι Γερμανία και η Αυστρία περί διαφορετικό ε, για την κατάρτιση των νέων, για την επαγγελματική επιμόρφωση, για την εμπλοκή των επιχειρήσεων της βιομηχανίας αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε από πλευρά των δημοσίων αρχών να βελτιώσουμε την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων και σε αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ανάγκη για ε, χρονικά περιθώρια μεταξύ των συστάσεων αναχώρα και της υιοθέτησή τους από το Συμβούλιο, όπως ανέφερε και άλλος συνάδελφος. Αυτό θα ενισχύσει και το δημοκρατικό διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ ημών και ημών ε, από τις δύο πλευρές δηλαδή, των κοινοβουλίων, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις, τις που είναι, όπως είπα, ο στόχος το στόχο της ε, βελτίωσης της δράσης των δημοσίων αρχών, όπως είπε και η κυρία Νταμνίου, τα Πρέπει να κοιτάξουμε την χρήση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου του ευρωπαϊκού προπολογισμού, ώστε να, βελτι... να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ να βελτιώσουν τα συστήματά του, γιατί ω εκ τη φύσεω ε, η ε, καινοτομία αυτή, η ανανέωση καλύτερα, είναι δαπανηρή. Αν χρειάζεται νέα τεχνολογία για την ανανέωση του δημοσίου, του κρατικού γίγνεσθε, ασφαλώ και θα πρέπει να υποστηριχθούν οι χώρε που έχουν ανάγκη στο να προσαρμόσουν προ την κατεύθυνση αυτή τα συστήματα τη δημόσια διοίκηση. Αλλά επίση θα ήθελα να πω ότι το Fourth Pact, το Six Pact, το Two Pact, το Fiscal Compact, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν με μέτρα σκληρά για τους ε, συμπολίτε μου πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα ότι φέρνουν αποτέλεσμα και την εξυγένωση του προπολογισμού αλλά και την επίτευξη της ανάπτυξης. Εάν δεν επιτύχουμε την ανάπτυξη με επενδύσεις, με ε, θέσεις εργασίας δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τους πολίτες ό,τι και να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο εισηγητής για τις καταληκτικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Όχι μόνο εγώ ως εισηγητής αλλά και οι σκιώδη εισηγητές των λοιπόν ομάδων καταγράφουν με βέβαιο στις προτάσεις σας και στις επόμενες συζητήσεις θα δείτε ότι θα δοθεί ευκαιρία για την αναζήτηση συμβαστικών λύσεων. Δεν θα απαντήσω σε όλες τις παρατηρήσεις, μία μόνο ή δύο ε, προτάσεις για να κλείσουμε τη συζήτηση. Καταρχάς, πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε κομμάτι μιας νομισματικής ένωσης που είναι η Ευρωζώνη και η οποία συνεπάγεται υποχρεώσεις αλλά και προϋποθέσεις και νομίζω ότι υπόθηκε άλλωστε ότι όταν, δημιουργήθηκαν, όταν δημιουργήθηκε η Νομισματική Ένωση δεν είχαν τηρηθεί αυτές οι προϋποθέσεις και σε αυτό ακριβώς έχει αποτύχει το ε, σχέδιο. Χώρες οι οποίες μόνες τους έλεγχαν εάν τηρούν τους κανόνες, ήταν δηλαδή και δικαστής και δικαζόμενος στο ΣΥΠΗΝ, ε, απέδειξαν με τη συμπεριφορά αυτή ότι δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν μαζί με τα κράτη-μέλη τα ίδια θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ουδέτερος διαιτητής, κριτής στην υπόθεση αυτή να συμμετέχει. Μια διαδικασία που ήθελα να υπογραμμίσω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Ε, για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα ελλείμματα επίσης. Άκουσα τα σχόλια των συναδέλφων που αναφέρονται στις πολιτικές ε, λιτότητες, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είχαν ε, αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Φυσικά αυτό για ορισμένε χώρε μπορεί να κρίνεται και λόγω του σημείου κινήσεως, γιατί αν ως σημείο κινήσεως έχουμε την κρίση, τότε είναι τα πράγματα δύσκολα. Αλλά τα κράτη τα οποία θέλησαν λόγω της κρίσης να ε, κάνουν μια διόρθωση πορείας ή να υποστηριχθούν. Είδαν αποτελέσματα. Δεν μίλησε όμως ποτέ κανείς για το γιατί υπήρξαν τα προβλήματα, γιατί υπήρξαν τα ελλείμματα, γιατί κάποιες χώρες σε εποχή που μπορούσαν ακόμα έκαναν ε, τις μεταρρυθμίσεις τους όπως η Γερμανία, ενώ κάποια άλλα κράτη δεν το έπραξαν. Άρα λοιπόν έχουμε και τις μεταρρυθμίσεις και την μερική αυτή αιρεσιμότητα που είναι από την πλευρά του το κράτος κάνει τη δουλειά του, τα καθήκοντά του και από την άλλη παρακολουθείται και επαληθεύεται και συνοδεύεται αυτή η δουλειά. Και ένα τελευταίο σχόλιο, χρειάζεται τόντι να ξανασυνδέσουμε την ανταγωνιστικότητα με την ανάπτυξη, να δώσουμε προοπτικές, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και κυρίως των νέων και αυτό απαιτεί ασφαλώς ένα μείγμα μέτρων. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν οι παριθμόν τέσσερα περάγραφος της εκθέσεώς μου αλλά και η πέμπτη, κυρίως τέταρτη όμως, ιδιαιτέρως υπογραμμίζει όμως ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με βάση ε, το μισθολογικό κόστος η Ευρώπη, τις ε, ξένες αγορές. Θα χρειαστεί να υπογραμμίσουμε τον παράγοντα προϊόντα, καινοτομία, να αναστήσουμε νέε αγορέ. Αλλά βέβαια θα χρειαστούμε και επενδύσει ιδιωτικέ και δημόσιε και αυτό βεβαίω θα ε, έχει αποτελέσματα ανάλογα με το πώ θα γίνει. Έγινε μια αναφορά από του Βέλγου συναδέλφου για τον περιφερειακό τη Αμβέρσα με ένα μεγάλο προπολογισμό υποδομών. Με 85% όμω χρηματοδότησε τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι δημόσιο το χρήμα που τον χτίζει τον αυτοκινητόδρομο αυτόν. Άρα βλέπουμε ότι ο συνδυασμό του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να φέρει πολύ καλά και επωφελή αποτελέσματα. Επίση, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι κομμάτι για τη ε, δημοκρατική διαδικασία αλλά και την ε, αποδοχή των ε, συστάσεων ανακράτος που αναφέρθηκε επίσης με ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και τα, στα όσα είπε ο τελευταίος Πρέπει να προσέχουμε η διαδικασία που ακολουθούν τα κράτη-μέλη και υπενθυμίζω και το Six πακέτο και το και το Fiscal Compact ότι υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη-μέλη κατά μέλη με ε, ε, με εθελοντικό τρόπο. Το αποδέχθηκαν, πάση περιπτώσει, εκουσίω. Γι' αυτό λοιπόν τώρα πλέον καθήκον του είναι να κάνουν τι μεταρρυθμίσει των υποδεμών, να ε, καθοδηγήσουν τι επενδύσει, αλλά αυτό να, και, ταυτόχρονα και να λογίσουν τα οικονομικά του, ώστε να έχουμε σαν αποτέλεσμα την αντιμετώπιση τη ανεργία και κυρίω ε, τη ανεργία των νέων. Ε, όπως είπα όμω, χρειάζονται οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει, και πρέπει πάνω απ' όλα τα κράτη-μέλη να αντιληφθούν γιατί χρειάζονται αυτή τη μεταρρύθμιση. Τη χρειάζονται όχι για τι Βρυξέλλε, αλλά για να εξασφαλίσουν μια ανταγωνιστική οικονομία, μια αποτελεσματική οικονομία, μια οικονομία που να μπορεί να εξάγει και να δημιουργεί και πάλι πλούτο και ευημερία που χρειάζεται ο πολίτη, τη χρειάζεται τόσο όσο και την επιθυμεί. Ε, γι' αυτό λοιπόν και ευχαριστώ του συναδέλφου εδώ που ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα Εθνικά του ε, Κοινοβούλια. Ήταν επικοδομητική πολύ η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να σας δω σύντομα στην επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο Και τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω από πλευρά μου του συναδέλφου των Εθνικών Κοινοβουλίων για, τις πολύτιμες, για την πολύτιμη συνεισφορά τους στη συζήτηση. Η διαδικασία της ενίσχυσης της δημοκρατικής λογοδοσίας στην ε, διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι εν εξελίξη. Προχωρούμε, κάνουμε βήματα προόδου. Αυτή η συνάντηση ήταν πολύ καλή. Είχαμε πολύ καλές συνεισφορές και από σας, από τις προτάσεις σας και ελπίζουμε και για σας αυτή η συζήτηση να σας επιτρέψει να ε, διαδραματίσετε από πλευρά σας τον ρόλο σας πολύ πιο αποτελεσματικά, το σημαντικό αυτό ρόλο που έχετε στα εθνικά σας κοινοβούλια, ώστε να ε, συνδυάσετε ρόλους ε, νομοθεσία περί σταθεροποίησης και συστάσεις ανακράτους με το νομοθετικό σας έργο. Υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη, σημειώνω, τα εθνικά αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχουν το ταχύτερο, ε, δηλαδή σε πιο πρώιμο ε, στάδιο, αλλά και πιο αποτελεσματικά στην επεξεργασία των συστάσεων ανακράτος. Αυτό ισχύει, όπως είπα, για τα εθνικά όσο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτή τη γραμμή μπορούμε να συνεργαστούμε και πιστεύω μπορούμε να βρούμε λύσεις κοινή πορεία για να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομοποίηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η προσεχής μας ε, συνάντηση και για το χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένα για την έκθεση αυτή. 7 Οκτωβρίου έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια στην δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. Αυτά και ευχαριστώ πολύ.